Colleagues, I think it's time to start. We know that there are some petitioners. Συνάδελφοι, να ξεκινήσουμε. Ξέρουμε ότι έχονται κάποιοι αναφέροντες. Αλλά μια και περιμένουμε να δούμε τα τυπικά. Τα τυπικά σημαίνει η οθέτηση της υπηρεσίας διάταξη. 24 σημείο, 307 αναφορά θα συζητηθεί πριν από το σημείο 20. που αφορά του Βρετανού υπηκόου οι οποίοι διαμένουν σε άλλε χώρε μέλη. Το σημείο 22 θα συζητηθεί το απόγευμα και νομίζω ότι μετά από αυτά, αν συμφωνείτε και εσεί, μπορούμε να εγκρίνουμε την ημέρα διάταξη. Ευχαριστώ. Έχω κάποιε ανακοινώσει καταρχά, με χαρά υποδέχομαι την κυρία Φάνη Φροντέ, νέα συνάδελφο στην Γραμματεία, που έχει και από άλλες επιτροπές, η τελευταία ήταν περιβάλλοντος και επειδή έχουμε πολλά θέματα που αφορούν αυτό ακριβώς το πεδίο, αυτό το ζήτημα, νομίζω θα είναι πολύ χρήσιμο να σας έχουμε εδώ ως μέλος της γραμματείας. Είστε λοιπόν μια πολύ καλή ενίσχυση της Επιτροπής μας. Να την υποδεχτούμε, ε, ε, σηκωθείτε να σας δουν οι συνάδελφοι για να σας υποδεχτούμε. Καλώς ορίσατε λοιπόν και πάλι και ελπίζω όλοι να είναι καλοί μαζί σας. Επίσης να σας ενημερώσω ότι δεν θα έχουμε σήμερα το απόγευμα δανέζικη διερμηνία επειδή απλά και μόνο δεν υπάρχουν αρκετοί διερμηνείς στη διάθεση της υπηρεσίας για σήμερα το απόγευμα επειδή γίνονται πολλά παράγγλα και ιδιαίτερα η εκδήλωση του κ. Ταγιάννη υψηλό επίπεδο για τη μετανάστευση σήμερα το απόγευμα, οπότε δεν υπάρχουν απαραίτητε διερμηνεί. Ελπίζω όσοι χρειαστούν διερμηνία στη ιδανική γλώσσα να ακούσουν τα σουηδικά που μοιάζουν πάρα πολύ ούτω ή άλλως. Ξέρετε ότι δεν έχουμε τίποτα άλλο στα διάφορα σήμερα. Έχουμε όμω κάποια πολύ ενδιαφέροντα σημεία στην ημερήσια διάταξή μας. Και το πρώτο σημείο που θα συζητήσουμε είναι η παρουσίαση της μελέτης με θέμα αντίκτυπος του Brexit σε σχέση με το δικαίωμα υποβολής αναφορών καθώς και στις αρμοδιότητες, τις ευθύνε και τις δραστηριότητε της Επιτροπής Αναφορών. Η καθηγήτρια Ελενόρ Σπαβέντα είναι η συγγήτρια. Χαίρομαι που είστε εδώ, θα σας το λόγο αμέσω. Απλά και μόνο να σας υπενθυμίσω ότι εμείς στην Επιτροπή μας Από πέρσι έχουμε δεχτεί 140 αναφορές σε σχέση με το δημοψήφισμα του Brexit που έγινε πριν περίπου ένα χρόνο σε σχέση με τις επιπτώσεις από τις διαπραγματεύσεις που μόλις τώρα ξεκίνησαν τη Δευτέρα. Ποικίλουν αυτές οι αναφορές πάντως. Η μεγάλη πλειοψηφία όμως αυτών αναφορών αφορά θέματα πολιτών, θέματα ηθαγένειας. Θα ακούσουμε σήμερα λοιπόν τους αναφέροντες και θα κάνουμε συζήτηση. Νομίζω ότι έγκαιρα προσφέρουμε ή δίνουμε τη δυνατότητα για αυτό το φόρουμ συζήτησης μετά από αυτές τις διαπραγματεύσεις που μόλις ξεκίνησαν. Σήμερα λοιπόν έχουμε την Κομισιόν και την μόνιμη αντιπροσωπεία του Ηνωμένου Βασιλείου στην Επιτροπή μας που θα ακούσουν τις αναφορές αυτές και θα παρακολουθήσουν τη συζήτηση. Όλοι υποσχέθηκαν να μεταφέρουν τα μηνύματα στις αντίστοιχες διαπραγματευτικές ομάδες και σήμερα το απόγευμα θα ακούσουμε και τους εμπειρογνώμονες, θα δούμε επίσης και ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα του κ. Μπαρνιέ, του κυρίου Διαπραγματευτή εκ μέρου τη Ένωση, και μετά θα ακούσουμε τη συναδελφό μα την κυρία Ντανούτα Χιμπνερ που είναι στην Επιτροπή, στη Διεθνή Επιτροπή για το Brexit στο Κοινοβούλιο και είναι μέλο τη Επιτροπής ΑΦΕΤ. Μετά βέβαια θα πάμε στου αναφέροντε και θα ακούσουμε τι ανησυχίε και το περιεχόμενο των αναφορών του. όλη μέρα σήμερα και το απόγευμα. Αλλά Ας ξεκινήσουμε με αυτή την μελέτη που ανέθεσε η Επιτροπή μας, ένα πάρα πολύ χρήσιμο εγγραφό. Αυτό είναι, εδώ το βλέπετε, το οποίο συνιστώ σε όλους σας, είναι διαθέσιμο εδώ στην αίθουσα. Θα δώσω λοιπόν το λόγο τώρα στην εμπειρογνώμονά μας, την κυρία Ελεανόρ Σπαβέντα. Um, thank you very much Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση σήμερα και για την πρόσκληση να γράψουμε αυτήν την μελέτη. Όταν αρχίσαμε τη συγγραφή της μελέτης ήταν ως αντίδραση σε αναφορές που λάβαμε από ε, διάφορους ανθρώπους στην Επιτροπή Αναφορών που αφορούσαν το Brexit και η μελέτη λοιπόν εστιάζει στα εκλογικά δικαιώματα, το δικαίωμα στην αναφορά, τις πρωτοβουλίες πολιτών φυσικά, αλλά η πλειοψηφία ε, της, ε, μάλλον το κυριότερο μέρος της μελέτης ασχολείται με τα δικαιώματα των πολιτών. Ασχολείται με αναφορές οι οποίες ε, όταν αρχίσαμε τη συγγραφή της μελέτης ήταν το κύριο κομμάτι της. αφορούν την κατάσταση για τους πολίτες της του Ηνωμένου Βασιλείου που ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και των και για πολίτε τη Ένωση των 27 που ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και προσπαθήσαμε λοιπόν να εντοπίσουμε του κινδύνου που ε, αντιμετωπίζουν και τους κινδύνους για τα θεσμικά όργανα κατά τη ε, διάρκεια των διαπραγματεύσεων για το Brexit. Προσπαθούμε να εντοπίσουμε κάποιους τομείς ε, που οι πολίτες είναι πιο ευάλωτοι απέναντι στα γεγονότα. Ε, υπήρξαν ορισμένες αναφορές οι οποίες ανέφεραν ότι οι ε, πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση που ζουν πάνω από 15 χρονικοί δεν έχουν το δυνα... την δυνατότητα ψήφου και κάποιοι αναφέροντε ε, εξέφραζαν τη γενικότερη δυσαρέσκειά τους για την όλη διαδικασία. Ω αντίδραση σε όλα αυτά ε, υπάρχει ε, λοιπόν το πόρισμα της μελέτης. Η απόφαση όμως για εκλογικά δικαιώματα των ε, Βρετανών πολιτών και γενικότερα άλλων πολιτών είναι αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών. Τα θεσμικά όργανα λοιπόν δεν έχουν από τις συνθήκες κάποια εξουσία να ε, δράσουν. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχει κίνδυνος οι πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου που ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση να χάσουν το δικαίωμα να ψηφίζουν για... σε διάφορες εκλογές, σε ευρωεκλογές ας πούμε. Οι πολίτες της Ένωσης στο Ηνωμένο Βασίλειο θα ε, περάσουν από ένα καθεστώς ε, που διέπονται από το ευρωπαϊκό δίκαιο σε ένα άλλο καθεστώς που υπόκειται στο Βρετανικό. Δηλαδή, ένας πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορεί να ψηφίσει στον Ηνωμένο Βασίλειο για ε, ε, προεκλογέ μόνο εάν η νομοθεσία επιτρέπει να το κάνει, του Ηνωμένου Βασιλείου επιτρέπει να το κάνει αυτό από απόσταση. Τώρα, εξαρτάται τι θα γίνει με την Ιρλανδία. Εδώ οι πολίτε μπορεί ε, τη Ένωση που ζουν στο Ηνωμένο Βασιλείο μπορεί να χάσουν το δικαίωμα να ψηφίζουν στι τοπικέ εκλογέ, εκτό εάν το κράτο ε, διαμονή του χορηγήσει αυτό το δικαίωμα. Υπάρχει μια εξαίρεση Σύμφωνα με του τους υφιστάμενους διακανονισμούς, οι πολίτε του ΗΠΑ στην Ιρλανδία μπορούν να ψηφίσουν και στις τοπικές ε, και στις εθνικές και στις ευρωεκλογέ σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο της χώρας. Τώρα, σε ό,τι αφορά το δικαίωμα στην αναφορά των ε, διαμεσολαβητή και τις πρωτοβουλίες πολιτών. Θα δείτε εδώ διάφορες ε, διακυμάνσεις, ε, διαφορές στα δικαιώματα των ε, Βρετανών πολιτών. Συγκεκριμένα, οι Βρετανοί πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 θα διτηρήσουν το δικαίωμα στην αναφορά και το δικαίωμα προσφυγής στον Ευρωπαϊκό Μεσολαβητή, διότι αυτό είναι ένα δικαίωμα που χορηγείται σε όλους τους κατοίκους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα χάσουν όμως το δικαίωμα συμμετοχής στις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες πολιτών. Αυτό το δικαίωμα το έχουν μόνο οι Ευρωπαίοι πολίτες, πολίτες Ένωσης. Τώρα, οι πολίτες Ένωσης στο Ηνωμένο Βασίλειο θα διατηρήσουν όλα τους τα δικαιώματα, αλλά η αποτελεσματικότητα αυτών των δικαιωμάτων μπορεί να είναι μειωμένη. Εδώ υπάρχει ένα ερωτηματικό. Δεν γνωρίζουμε εάν τα αγγλικά θα παραμείνουν επίσημη γλώσσα και γλώσσα των συνθήκων μετά το Brexit. Αλλά ε, σε ό,τι αφορά την πρωτοβουλία πολιτών, να πω ότι οι περισσότερες πρωτοβουλίες γράφονται στα αγγλικά για προφανείς λόγους, γιατί χρειάζεται συμμετοχή από πολλά κράτη-μέλη για να ε, χαρακτηριστεί παραδέκτη. Υπάρχει λοιπόν ε, κίνδυνος ε, για το μέλλον και την αποτελεσματικότητα της πρωτοβουλίας των πολιτών και τη χρήση της αγγλικής ως γλώσσας επικοινωνίας. Όπως είπα, το κύριο κομμάτι της μελέτης αυτής αφορά τα δικαιώματα των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ένωση των 27 και των πολιτών της Ένωσης των 27 στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν προσπαθούμε εδώ να κάνουμε κάποια συγκεκριμένη πρόταση, να υποδείξουμε τι πρέπει να γίνει. Αυτό φυσικά είναι ε, θέμα των ε, διαπραγματεύσεων, αλλά προσπαθούμε να εντοπίσουμε και ίσως να ε, ρίξουμε φως στους κινδύνους που υφέρπουν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την ατζέντα των διαπραγματεύσεων, είναι ανοιχτή σε προσβάσιμη με όλου του πολίτες, είναι πολύ περιεκτική και προσπαθεί να διατηρήσει όσο το δυνατόν περισσότερο τα δικαιώματα όλων των ε, πολιτών ε, που, έχουν, ε, που διαμένουν εκεί. Τώρα, τη Δευτέρα θα δημοσιεύσει και το Ηνωμένο Βασίλειο την αντίστοιχη ε, εγκύκλιο. Τώρα, μετά το Brexit, τι θα γίνει. Ε, σύμφωνα με το Βρετανικό Δίκαιο υπάρχουν διάφορα είδη ε, πολιτών. Υπάρχουν οι πολίτες που διαμένουν για λίγο, άδεια βραχίας παραμονής, 0 έως 3 μήνες. Εδώ δεν γνωρίζουμε τι θα γίνει, δεν γνωρίζουμε αν θα υπάρξει κάποια συμφωνία για ελεύθερη ε, κυκλοφορία των πολιτών ε, χωρίς απέτηση θεώρησης. Μετά, οι μεσοκάτοικοι που είναι η πιο ευάλωτη ομάδα είναι οι, πολίτη, οι πολίτες οι οποίοι μένουν στο Ηνωμένο Βασίλειο από τρεις μήνες έως πέντε χρόνια. Αυτή η μέση παραμονή. Αυτό εδώ είναι μια περίπτωση η οποία δίπεται από πολλές προϋποθέσεις. Και μετά Υπάρχουν και οι μόνιμοι κάτοικοι. Ένας πολίτης που μένει πάνω από πέντε χρόνια σε ένα κράτος μέλος θεωρείται μόνιμος κάτοικος. Υπάρχουν και εδώ ε, ορισμένες προϋποθέσεις οι οποίες όμως δεν, χρειάζεται να, ε, δεν υφίστανται μετά από πέντε χρόνια διαμονής. Ας αρχίσουμε τώρα τονίζοντας και σκιαγραφώντας τα εφιστάμενα δικαιώματα των ε, πολιτών της Ένωσης που μένουν εκτός. Κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας, κατοικίας και ίσης μεταχείρισης. Δεν μπορούν λοιπόν να υφίστανται διακρίσεις βάσει εθνικότητας για κανένα ζήτημα. Οι πολίτες επίσης έχουν δικαιώματα οικογενειακής επανένωσης, τα οποία είναι πολύ πιο γενναιόδωρα από ό,τι προβλέπει το εθνικό δίκαιο. Εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο αυτό είναι πολύ έντονο. Τα δικαιώματα οικογενειακής επανένωσης είναι πολύ πιο περιορισμένα από εκείνα που δίνει το ευρωπαϊκό δίκαιο. Υπάρχει το δικαίωμα να επιστρέψουν στο κράτος μέλος προέλευσης και να πάρουν μαζί τους τις οικογένειές τους αφού μετακομίσουν εκεί και αυτό θα μας απασχολήσει στο μέλλον διότι υπάρχει ο κίνδυνος Βρετανοί πολίτες που ε, μετακόμισαν, μετανάστευσαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 και θέλουν να επιστρέψουν, τώρα ε, ενδέχεται να υπόκεινται στην εθνική νομοθεσία και όχι στην ευρωπαϊκή. Οι Ευρωπαίοι πολίτες επίσης ε, χαίρουν εκτεταμένης προστασίας από απέλαση, όμως τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας μας λένε ότι αυτό δεν εφαρμόζεται. Υπάρχουν συγκεκριμένες, πολύ περιορισμένες στον αριθμό περιπτώσεις, κατά τις οποίες έχουμε δει πως η ευρωπαϊκή θα είναι της Ένωσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναντίον του πολίτη. Μετά. Πώς λειτουργεί τώρα εδώ το ευρωπαϊκό δικείο. Θα σας τα πω πολύ απλά, απλοποιημένα. Βασικά, για να μπορεί ένας πολίτης να διαμένει σε ένα κράτος μέλος διαφορετικό από εκείνο της επικότητάς του πρέπει να πληρεί κάποιες προϋποθέσεις. Πρέπει να είναι είτε οικονομικά ενεργός ο πολίτης είτε οικονομικά ανεξάρτητος. Οικονομικά ενεργός. Είναι ένας πολίτης που είτε είναι εργαζόμενος είτε ε, αυτοαπασχολούμενος. Ένας εργαζόμενος ε, κατά το ευρωπαϊκό δίκαιο είναι ε, ε, οποιοδήποτε ασκεί κάποια ανεμπόδιστη δραστηριότητα ε, με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Είτε είναι η μία απασχόληση, αλλά καλύπτονται και ακόμα εκείνοι που δουλεύουν ελάχιστε ώρε, δύο-τρει ώρε. Αυτέ είναι περιπτώσει που το δικαστήριο τις έχει δεχτεί έτσι ώστε οι πολίτε να απολαμβάνουν την ε, προστασία ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα, θα αναφερθώ και αργότερα σε αυτό, αλλά υπάρχουν ορισμένοι που έχουν άτυπη σχέση εργασία ή μια απασχόληση, ώρα, συμβόλαια ε, μηδενικών ορών, οι οποίοι κινδυνεύουν με τον Brexit. Ακριβώς γιατί γνωρίζουμε πως υπάρχουν κάποια ε, αρκετά κρατημέλη που δεν αναγνωρίζουν ακόμα και σήμερα τις αποφάσεις του δικαστηρίου και δεν τις εφαρμόζουν. Τώρα δεν υπάρχουν ελάχιστες απαιτήσεις ε, στο ευρωπαϊκό δίκαιο και σε ό,τι αφορά τους αυτοαπασχολούμενους υπάρχει τώρα ένα ε, κατώτατο ε, κατόφλι κεφαλαίο. Δηλαδή, κανένα συνδραυλικό που πηγαίνει από το Ηνωμένο Βασίλειο στη Γαλλία δεν θα πρέπει να δείξει ότι έχει ένα ελάχιστο ε, τζίρο, ένα ελάχιστο κύκλο εργασιών κάθε χρόνο. Αυτοί οι πολίτες τώρα, οι οποίοι είναι οικονομικά ενεργοί, στην ουσία απολαμβάνουν ε, τα πλήρη δικαιώματά τους. Η μεταχείριση, ε, πρόσβαση στις υπηρεσίες του κράτους μέλους, ακόμα και αν δουλεύουν σε καθεστώς απασχόληση ή δουλεύουν λιγότερες ώρες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τις γυναίκες οι οποίες ε, φροντίζουν μέλη της οικογένειας. Τώρα, οι ανεξάρτητοι πολίτες, για παράδειγμα, συνταξιούχοι, φοιτητές, μη ενεργοί οικονομικά πολίτες. Αυτοί έχουν δικαίωμα διαμονής σε οποιοδήποτε κράτος μέλος της Ένωσης. Αυτοί οι πολίτες πρέπει να έχουν επαρκείς πόρους και ε, να έχουν κάποια ε, ασφάλιση γενομικής περίθαλψης. Συμπεριλαμβάνονται φοιτητέ εδώ και, πολύ σημαντικό για τους Βρετανούς πολίτες στο εξωτερικό, οι συνταξιούχοι. Και ε, υπό τον αισθενισμό του ασφαλιστικού συστήματος ισχύουν τα εξή. Δεν χρειάζεται ο Βρετανός πολίτης να έχει κάποιο πρόγραμμα ασφάλισης γιατί αυτό το καλύπτουν τα κράτη-μέλη. Οι συνταξιούχοι όμως εδώ ε, έχουν μεγαλύτερες δυσκολίες στο να ασφαλιστούν. Σε αυτό το στάδιο τώρα βλέπουμε ότι πολλοί πολίτες της Ένωσης δεν γνωρίζουν ότι το δικαίωμα κατοικίας, ε, νόμιμης κατοικίας ε, συνεπάγεται και να είναι ασφαλισμένοι. Αυτό γιατί οι περισσότεροι πολίτες της Ένωσης δεν ε, μεταναστεύουν σε κάποιο άλλο κράτος μέλος για να λαμβάνουν επιδόματα και αυτές οι προϋποθέσεις ε, και αυτό, αυτές, ε, αυτές λοιπόν οι προϋποθέσεις ε, ισχύουν ή τις μαθαίνουν οι πολίτες μόνο όταν ζητήσουν κάποιο πίδωμα. Αυτό λοιπόν πιστεύω πως είναι ένας τομέας που πρέπει να προσέξουμε πολύ. Τώρα, να εξετάσουμε εν συντομία το καθεστώς των Βρετανών πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μετά ε, το καθεστώ των Ευρωπαίων πολιτών στο Ηνωμένο Βασίλειο. Επέλεξα αυτή τη σειρά όχι επειδή υποτιμώ την, ε, τα προβλήματα που θα αντιμετωπίσουν οι Ευρωπαίοι πολίτες στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά διότι είναι μια περίεργη περίπτωση, είναι κάπως διαφορετικά τα πράγματα. Ε, μιλάμε και για βρετανικό δίκαιο και για ευρωπαϊκό. Υπάρχει μια σάφια στο τι θα ε, υπερισχύσει μετά το Brexit. Στη μελέτη λοιπόν... Ε, καταρχάς βλέπουμε ότι, υπάρχει ένα, ότι δεν υπάρχει προηγούμενο, δεν υπάρχει νομολογία, δεν υπάρχει κανένα πλαίσιο που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να μας καθοδηγήσει. Δύο, οι επιλογές, δύο πιθανότητες. Οι Βρετανοί πολίτες οι οποίοι έχουν αλλάξει χώρα καλή την πίστη θα ασκούν δικαιώματα που τους παρέχονται από το ευρωπαϊκό δίκαιο. Ξαφνικά λοιπόν αυτοί οι πολίτες, ξαφνικά μετά από κάποια διαδικασία θα διαπιστώσουν ότι δεν προστατεύονται. Και αυτοί οι Βρετανοί πολίτες μπορεί να επίπτουν σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις. Η μία να τους δούμε ως πρώην πολίτες της Ένωσης, δηλαδή να υπάρχει ένα προηγούμενο, να είναι άτομα που ήταν κάποτε πολίτες της Ένωσης, να τους δούμε δηλαδή με αυτό το καθεστώς και μια άλλη πρόταση, ε, εκείνοι οι άνθρωποι από τη μια μέρα στην άλλη να γίνουν υπήκοοι της χώρας. Και αυτή η θέση είναι πολύ πιο άσχημοι από το να θεωρούνται πρώην πολίτες της Ένωσης. Θα μπω σε νομικές λεπτομέρειες αργότερα ή δεν θα μπω μάλλον ιδιαίτερα σε λεπτομέρειες, αλλά να σας πω ότι οι Βρετανοί πολίτες στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχουν τη δυνατότητα να διατηρήσουν ε, τα δικαιώματα που απορρέουν από την Οδηγία 2038. Θα προσπαθήσω τώρα να τονίσω γιατί είναι τόσο ε, σημαντικό αυτό. Εδώ στη μελέτη θα βρείτε και έναν πίνακα που απαριθμεί τις διαφορές που θα προκύψουν ανάλογα με το πώς θα κατατάξουμε τους πολίτες μετά τον Brexit. Για τους Βρετανούς, επειδή κάποιοι αν έχουν ένα ιδιαίτερο καθεστώς θα διατηρήσουν το δικαίωμα διαμονής, εργασίας, δικαίωμα να είναι αυταπασχολουμένοι. Δεν θα υπάρξουν δηλαδή κάποιες προϋποθέσεις που θα τους επιβληθούν, αλλά θα συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν την πρόκληση ως φοιτητέ ή συνταξιδοτούμενοι. Και για το δικαίωμα των συνταξιούχων να μετακινηθούν και να διαμείνουν, αυτό θα πρέπει να συνοδευτεί από ένα συντονισμό όσον αφορά τα συστήματα κοινωνική πρόνοια. Και αν δεν υπάρχει αυτό ο συντονισμό, ο συνταξιούχο δεν θα καλύπτεται από το Εθνικό Σύστημα Υγεία τη Αγγλία. Και για του φοιτητέ έχουμε προβλήματα, επειδή οι περισσότεροι φοιτητέ, να σα πω ότι εγώ διδάσκω στο Πανεπιστήμιο, αγνοούν την ανάγκη για πλήρη ιατρική κάλυψη. Διαμένουν σε μια χώρα μέλος, αλλά δεν χρειάζονται προς το παρόν ιατρική κάλυψη. Αυτό δεν είναι ίσως πρόβλημα για τους προπτυχιακούς, αλλά για τους μεταπτυχιακούς υπάρχει πρόβλημα, γιατί καμιά φορά θέλουν να εγκατασταθούν στη χώρα στην οποία φοιτούν. και βέβαια οι Βρετανοί φοιτητέ θα διατηρήσουν το δικαίωμα για ίση μεταχείριση και βεβαίω θα έχουμε και την κάρτα διαμονής που αυτή τη στιγμή ε, δίδουμε σε ε, υποψηφίους ε, προς διαμονή από τρίτες χώρες. Με ναι, αυτή θα μπορούσαν να ταξιδέψουν και μετακινηθούν σε όλη την Ευρώπη. Αν αποφασίσουμε τώρα και όπως είπα προηγουμένω, εγώ μελέτησα αυτό το θέμα της ηθαγένειας, οπότε αν το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφασίσει διαφορετικά και τους χαρακτηρίσει ως υπηκόους τρίτων χωρών, ξαφνικά και άμεσα, χάνουν το καθεστώς που τους δόθηκε από τις συνθήκες. Οπότε η κατάσταση δεν είναι διατρά Επειδή ως Βρετανοί υπήκοοι θα υπόκεινται σε διαφορετικού κανόνες μετανάστευση σε όλε τι χώρε μέλη και υπάρχει ένα ερωτηματικό εδώ για την ε, Ιρλανδία, αλλά τέλος πάντων το λέμε στο τέλος τη ε, μελέτη, ότι μπορεί να υπόκειται σε υποχρεώσει θεώρηση, ε, ελάχιστε προποθέσει. Οι ανειδίκευτοι μπορεί να αντιμετωπίζουν ιδιαίτερο κίνδυνο, όπως αυτή με τα zero hours, αυτές τις συμβάσει εργασία. Και σε κάποιες Χώρε μέλη, ίσως ένας αυτοαποσχολούμενο μπορεί να μην λάβει καθόλου θεώρηση εκτό και να είναι πολύ πλούσιοι και το δικαίωμα τη μεταχείρισης θα εξαρτάται απολύτω από τι εθνικέ νομοθεσίε, δεν θα υπάρχει δηλαδή προστασία. Και να θυμάστε ότι αυτοί οι άνθρωποι μετακινήθηκαν ω πολίτε τη Ένωση. Δεν είναι άνθρωποι που μετακινήθηκαν μετά το Brexit. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει να προστατευτούν, γιατί η Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια περί αυτού πρόκειται. Ίσως λοιπόν μετά να υπόκεινται και σε υποχρεώσεις θεώρησης ε, στα πλαίσια της Σέγγεν, κάτι το οποίο θα πρέπει να είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης και μετά από πέντε χρόνια νόμις διαμονής θα μεταβούν στο καθεστώς των μακροχρονίων δεμενών των υπηκών τρίτων χωρών. Αλλά βέβαια αυτό δεν είναι τόσο ευνοϊκό όσο το καθεστώ το καθεστώς της Ένωσης για εμπικός χωρομελών της Ένωσης. Ό,τι και να γίνει λοιπόν, θεωρώ ότι υπάρχουν ιδιαίτεροι κίνδυνοι για αυτούς τους πολίτες και μάλιστα συστάσεις αυτές αφορούν όλους τους πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης στον Ηνωμένο Βασίλειο. Καταρχάς, όσον αφορά την προοπτική της Ιθαγένειας και το οποίο αυτό ξεκάθαρα η Κομισιόν, εδώ έχουμε να κάνουμε οποιαδήποτε μορφή μετανάστευση, μετακίνηση πριν από τη συμφωνία την οριστική στην οποία θα καταλήξουμε. Εδώ γίνεται λόγος ε, βέβαια για το άρθρο 50 αλλά από την σκοπιά του κοινωνικού δικαίου είναι δύσκολο να τεκμηριωθεί αυτό. Επίσης, αυτό που πρέπει να κάνουν τα θεσμικά όργανα είναι να καθορίσουν ξεκάθαρα τι εννοούν με τον όρο εργαζόμενος. Και αυτό επειδή σε μια άλλη μελέτη που κάναμε για την Γενική Διεύθυνση Απασχόληση τη Κομισιόν είδαμε ότι σε πολλέ χώρε μέλη δεν δεν ακολουθούνται οι κατευθυντήριες γραμμές για το καθεστώς των εργαζομένων που αποφάσισε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Και ιδιαίτερα πολλές χώρες μέλη αρνούνται να παραχωρήσουν αυτό το καθεστώς εργαζόμενου σε όσους εργάζονται με συμβόλαιο μηδενικών ωρών ή σε μερική απασχόληση. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε τι γίνεται τώρα υπό του όρου του Brexit, γιατί αν δεν αναγνωρίζεται το καθεστώς των μερικώς απασχολημένων, των ατύπων εργαζομένων, των εργαζομένων με μηδενικές ώρες, αν λοιπόν όλοι αυτοί δεν έχουν κάποιο καθεστώ μετά το Brexit θα χάσουν οτιδήποτε καθεστώ έχουν. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό γιατί ήδη είναι αρκετά σοβαρό αυτό που γίνεται από τώρα στο εσωτερικό των χωρών μελών. Αλλά ε, να θυμάστε ότι αν ένας πολίτης έχει πάει σε άλλη χώρα μέλο και δεν τους θεωρούμε εργαζόμενους κατά τη στιγμή του Brexit, τότε δεν θα έχουν κανένα απολύτω δικαίωμα υπό την ε, Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Οπότε εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία μπορείτε να διατηρήσετε το καθεστώς του εργαζομένου αν είστε άνεργος. Αλλά για να διατηρήσετε αυτό το καθεστώς θα πρέπει βεβαίως να καταγραφείτε στις, ε, στους κατατόπους ΟΑΕΔ. Αρκετοί πολίτες το γνωρίζουν αυτό, αλλά πολλοί όχι γιατί μπορείτε ας πούμε, να δουλεύετε μέχρι τον Ιούνιο, να πάτε διακοπές και από το Σεπτέμβριο να ξαναψάξετε για δουλειά, αλλά δεν μπορείτε να λάβετε επίδομα Οπότε θεωρώ ότι είναι κρίσιμη σημασία η έλλειψη καταγραφής ή η μη καταγραφή στις ε, δομές, στις υπηρεσίες ανεργίας να μην επηρεάζει ακριβώς το δικαίωμα για επιδόματα ανεργίας. Γιατί σε αυτή την περίπτωση τιμωρούμε τους ενάρετους ή τους τυχερούς που μπορεί να, έχουν, να διαθέτουν αρκετούς πόρους και μπαινοβγαίνουν στην απασχόληση. Γιατί αυτή είναι και η μορφή οικονομίας την οποία βλέπουμε να επικρατεί αυτή τη στιγμή. Οπότε η ευθύνη θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Αυτή τη στιγμή αν α πούμε είστε κάποιος που φροντίζει παιδιά, ηλικιωμένου, άτομα με αναπηρία, μπορεί να δείτε ότι το καθεστώς αυτό του εργαζομένου που έχετε διακόπτεται. Και αυτό θα ήταν βεβαίω ε, αρνητικό, γιατί με αυτόν τον τρόπο αφαιρεί ακριβώς ε, το καθεστώς αυτός μετά τον Brexit και βεβαίως ε, είναι και θέμα φύλου, γιατί περισσότεροι, τα περισσότερα από αυτά τα άτομα είναι γυναίκες. Θεωρώ λοιπόν ότι κατά την άποψή μου αυτή η έλλειψη η ιατρικής κάλυψης θα πρέπει να διαδραματίζει κάποιο ρόλο αναδρομικά. Γιατί έχουμε αυτή την Ευρωπαϊκή Κάρτα Υγείας, έχουμε την ελεύθερη κυκλοφορία, έχουμε την Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια και νομίζω ότι έχουμε δημιουργήσει προσδοκίες στους πολίτες ότι αυτό δεν το χρειάζονται. Οπότε θα έλεγα ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί για να μην τιμωρήσουμε, να μην ζημιώσουμε αυτούς τους ε, πολίτες που καλή την πίστη έδρασαν και δεν τήρησαν αυτές τις προϋποθέσεις. Και όπως είπε και η Κομισιόν και διευκρίνησε, προτίθεται να προστατεύσει τα μέλη των οικογενειών των, πολιτών των χωρομελων τη της Αν εσείς λοιπόν εσείς είστε πατριμένος με υπήκο της χώρας ή με ένα άτομο το οποίο είναι οικονομικά ενεργό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να διευκρινιστεί. Και βεβαίως εδώ μπλέκονται και παιδιά και το συμφέρον των παιδιών, ιδιαίτερα το δικαίωμα για εκπαίδευση που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη αυτές τις συμφωνίες. Επίσης θα πρέπει να υπάρξει, θα υπάρξει μάλλον ένα τεράστιο πρόβλημα και ήδη το βλέπουμε στο Ηνωμένο Βασίλειο με τις άδειε διαμονής σε σχέση με τα αποδεκτικά στοιχεία τα οποία απαιτούνται από πολίτες για να αποδείξουν ακριβώς το καθεστώς στο οποίο βρίσκονται. Και πάλι, εμείς είμαστε τυχεροί. Έχουμε δουλειά. Εγώ έχω, ας πούμε, τους φακέλους με τα προσωπικά στοιχεία ε, στους υπολογιστές ε, για την εφορία κλπ. Αλλά αυτό δεν ισχύει με όλους τους πολίτες, οπότε θα πρέπει να προσέξουμε με τα αποδεικτικά στοιχεία και το είδο αποδεικτικών στοιχείων που θα ζητήσουμε από του πολίτε. Βεβαίω όλα αυτά θα πρέπει να είναι ενιαία και στι 27 χώρε μέλη. χωρί δηλαδή να υπάρχει περιθώριο διακριτική ευχέρεια στι χωρε μέλη, γιατί ξέρουμε ότι κάποιε ε, χωρε μέλη είναι πιο αποτελεσματικέ, άλλε χώρε μέλη είναι λιγότερο αποτελεσματικέ. Και ό,τι και να αποφασίσουμε σε σχέση με τα αποδεικτικά αυτά στοιχεία θα πρέπει να επιτρέπουμε στους πολίτες να αποδείξουν την κατάστασή τους στο καθεστώς στο οποίο βρίσκονται με οποιοδήποτε τρόπο, έστω και αν αυτό δεν προβλέπεται. Και αυτό θα πρέπει να το βάλουμε κάπου στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Τώρα, τι συμβαίνει στους ε, Ευρωπαίους πολίτες ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ε, τη απουσία συμφωνίας αυτό το τονίζω, ελπίζω να μην ε, φτάσουμε εκεί. Το Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκεται σε δύσκολη θέση και εγώ μιλώ ως κάποια η οποία εργάζεται σε κάποιο πανεπιστήμιο και τα Βρετανικά πανεπιστήμια απασχολούν πολλούς από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μεταξύ αυτών και εμένα. Θα μπορούσε το Ηνωμένο Βασίλειο να αποφασίσει να μας δώσει αυτομάτως μια εργασίας. Αυτό μπορεί να λειτουργήσει ή όχι. Το πρόβλημα είναι ότι θα μπορούσε να λειτουργήσει μια χαρά για άτομα σαν και εμένα που έχουν ε, μόνιμη σύμβαση απασχόλησης και να είναι πολύ πιο δύσκολη η κατάσταση για όσους έχουν ε, προσωρινή απασχόληση ε, και δεν θα λειτουργεί σύμφωνα με το τωρινό μεταναστευτικό δίκαιο για όσους δουλεύουν part-time ή είναι ορομίστη ή έχουν κάποια μη συνήθι μορφή εργασία. Ε, που ξέρουμε παραδείγματο χάρη στον χώρο τη εστίαση ότι είναι πολύ συχνέ αυτέ οι συμβάσει. Επίση υπάρχει το θέμα του χρονισμού γιατί αυτή τη στιγμή οι αρχές του ΕΒ αναγνωρίζουν το καθεστώς του εργαζομένου μετά από τρεις μήνες απασχόλησης που και πάλι βάζει τα άτομα εκείνα τα οποία είναι σε ασυνήθη κατάσταση ή του ορομίστιους σε πολύ ευπαθή κατάσταση. Αυτή τη στιγμή για την αυτοαπασχόληση έχουμε την ελάχιστη επένδυση 50.000 λιρών και την ελάχιστη απέτηση αποταμίευσης και αν ισχύσει αυτό για τους πολίτες της Ένωσης τότε ο περίφημος πόλωνος υδραυλικός μάλλον θα ε, βρεθεί εκτός ε, Ηνωμένου Βασιλείου δεν θα έχει δικαίωμα να παραμείνει. Οι οικονομικά ανενεργοί όπως πάντα ε, είναι πολύ ευάλωτοι, χρειάζονται κάποιο ελάχιστο εισόδημα και επίσης και αυτοί θα έχουν ε, σοβαρό κίνδυνο. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, μην ξεχνάμε, υπάρχουν πολύ ακριβά τέλη για την αίτηση βίζας ε, και αυτό επίσης ε, είναι κάτι το ανησυχητικό. Επίσης ε, για τα μέλη της οικογένειας η κατάσταση θα είναι καταστροφική γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει μια ελάχιστη απέτηση εισοδήματο για τα μέλη της οικογένειας που είναι πολύ υψηλή, είναι πάνω δηλαδή από το βασικό μισθό. Είναι γύρω στις 18.600 λίρες, οπότε πολλές ε, νοσοκόμες ε, παραδείγματος χάρη ε, δεν θα έχουν τον δικαίωμα να έχουν την οικογένειά τους κάτι το οποίο δεν νομίζω ότι είναι ιδεώδης λύση οπότε ξέρετε ότι εντάξει δεν θα κάνω εγώ συστάσεις ή τα θεσμικά όργανα για το πώς θα πρέπει να κινηθεί το Ηνωμένο Βασίλειο αλλά η σύστασή μου αφορούν περισσότερο τα το τι πρέπει να κοιτάξετε στις διαπραγματεύσεις, δηλαδή αυτά δεν θα πρέπει να ισχύσουν ούτε ως υποθέσεις για το μη ελάχιστο εισόδημα και τις ώρες εργασίας. Υπάρχουν α, αυτές οι απαιτήσει στο ΕΒ. Βασίλειο. Μπο, ε, μπορεί να τα αντικρούσει κάποιος, αλλά πολλοί εργαζόμενοι να μην ξέρουν ότι έχουν αυτό το δικαίωμα. Να λάβουν μία επιστολή και να θεωρήσουν ότι αυτό ήταν και πρέπει να φύγουν. Πρέπει λοιπόν να ξεκαθαρίσουμε ότι μπορεί να επιβληθούν απαιτήσει εισοδήματος και ωρών εργασίας. Ε, και το ίδιο και για τους ε, αυτοαπασχολούμενους. Και... Στο Ηνωμένο Βασίλειο αυτή τη ε, στιγμή τα στοιχεία τα οποία πρέπει να δώσει ο εργαζόμενος είναι τεράστια, 80 σελίδες έγγραφα και ε, δεν ξέρουμε και πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις. Πρέπει μετά το Brexit λοιπόν για τα άτομα τα οποία βρίσκονται στο Ηνωμένο Βασίλειο να μειωθούν οι απαιτήσει των πραγμάτων που πρέπει να αποδείξουν ε, τα, τα άτομα στο ελάχιστο. Και μπορεί να το θέλει και η Βρετανική κυβέρνηση, γιατί το να επεξεργαστούν αιτήσει ε, τριών εκατομμυρίων ατόμων με τη μία δεν είναι εύκολο. Οπότε ε, νομίζω ότι, όπως είπα, και τα οικονομικά ανενεργά άτομα δεν θα πρέπει να τιμωρηθούν επειδή δεν, έχουν, δεν είχαν ασφάλεια υγεία στο παρελθόν. Και υπάρχει και το ζήτημα του Ηνωμένου Βασιλείου όπου ο Επίτροπος είπε ότι η πρόσβαση στο NHS είναι ασφάλιση υγείας. Είναι ένα ζήτημα ανοιχτό. Αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι ότι θα πρέπει να επιτρέψουμε στους οικονομικά ανενεργούς να πληρώσουν το τέλος το λεγόμενο υγείας που είναι πολύ χαμηλότερο από την ασφάλιση υγείας, είναι 150 λίρες. Ε, επίσης, το, ε, όταν πήγαν εκεί οι πολίτες ε, της Ένωσης, ήταν πολίτες της Ένωσης, υπαθόκαστος πήγαν Δεν δέχομαι ότι δεν είναι ευθύνη της Ένωση. Τώρα, λίγα λόγια για την μόνιμη κατοικία. Η μόνιμη κατοικία δίδεται μετά από πέντε χρόνια νόμιμης παραμονής το πρόβλημα είναι τώρα εδώ πέρα ότι το ΔΕΚ έχει ξεκαθαρίσει ότι η νόμιμη παραμονή είναι αυτή η οποία είναι σύμφωνη με την οδηγία 2004-38, δηλαδή οι πολίτες εάν είναι οικονομικά ανενεργοί πρέπει να αποδείξουν ότι είχαν οικονομική δραστηριότητα ή ασφάλιση υγείας, δηλαδή επαρκής πόρους και συνέχεια μια ε, συνεχή παρουσία. Δηλαδή επιτρέπεται ε, να είναι κανείς, ε, να απουσιάζει μόνο έξι μήνες το χρόνο ή πρέπει να είναι παρόν έξι μήνες το χρόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και υπάρχουν και άλλα προβλήματα ε, επίσης για την απόδειξη αυτού του πράγματος. Θεωρώ ότι ο σημαντικότερος κίνδυνος που έχουμε εδώ είναι η απόδειξη και η έλλειψη ενημέρωσης των πολιτών της Ένωση μετακόμισαν καλή την πίστη στο Ηνωμένο Βασίλειο για τους όρου που πρέπει να πληρούν και το πώ θα το αποδείξουν. Και πάλι, η δυνατότητα, παραδείγμα, το να μην έχει γραφτεί κανείς στο Ταμείο ανεργία ε, σημαίνει ότι δεν ε, κατοικεί. Και μπορεί να μην το ξέρουν αυτό. Λοιπόν, συστάσεις. Ε, τώρα. Πρέπει να σκεφτούμε ότι ο χρόνος και μόνο μπορεί να παρέχει ένα καθεστώς παραμονής μετά το Brexit, δηλαδή πέντε χρόνια ακόμα και αν δεν πληρεί κάποιος όρους, αλλά αυτό είναι αισιόδοξο νομίζω δεν θα συμβεί. Αλλά νομίζω πρέπει να αποφευθούν κάποιοι κίνδυνοι με την συμφωνία, δηλαδή το να μην έχει κανείς πάει στο Ταμείο Ενεργείας. Ότι θα πρέπει να υπάρχει μία σορευτική προσέγγιση στις περιόδους απασχόλησης. Δηλαδή αν κάποιος σταμάτησε να δουλεύει για να πάει διακοπές ή για να φροντίσει κάποιο άτομο, να υπάρχει, να ε, αντιμετωπίζεται συνολικά ο χρόνος. Πρέπει όμως να προσέχουμε ότι η φροντίδα ατόμων να μην διακόπτει ποτέ την κατοικία. υπάρχει ζήτημα διάκρισης ε, με βάση το φύλλο και να μην επιβληθεί αναδρομικά η συνολική ασφαλιστική Λοιπόν, θα σταματήσω εδώ. Τα υπόλοιπα τώρα σας λέω πώς θα ήταν τα πράγματα χωρίς συμφωνία. Πόσο άσχημα θα ήταν τα πράγματα. Υπάρχουν λοιπόν πίνακες σε ολόκληρη αυτή την ε, μελέτη. Και σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε σήμερα. Ελπίζω να μείνετε για να απαντήσετε σε ερωτήσεις των συναδέλφων. Ε, όμως ήδη δεν μας φτάνει ο χρόνος, έχουμε πολλούς αναφέροντες περιμένουν να πάρουν το λόγο, αλλά και την ε, συναδελφό μου εδώ, την κυρία Χούμπνερ, θα ήθελα όμως τώρα να σας παρουσιάσω τον επικεφαλής διαπραγμάτευσης, τον ε, Μισελ Μπαρνιέ, ο οποίος δεν μπόρεσε να έρθει σήμερα εδώ, αλλά έχει στείλει ένα μήνυμα για τους αναφέροντες που βρίσκονται στην αίθουσα. Ας ακούσουμε λοιπόν τον Μισελ Μπαρνιέ. Dear members of the Petition Committee, dear Cecilia, ladies and gentlemen, it is my pleasure to talk to you today even though I cannot be with you. Citizen first,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 Θα δώσω τώρα το λόγο στην Τανούτα Χούμπνερ, η είναι πρόεδρος της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων, η οποία είναι η καθήλυνα αρμόδια επιτροπή για ε, το θέμα της αποχώρησης του ΕΒ από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κυρία Χούμπνερ παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και είναι ε, μέλος της ε, Επιτροπής του Κοινοβουλίου για τον Brexit. Έχετε το λόγο σας. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα καταρχάς να σας ευχαριστήσω που μου δίνετε την ευκαιρία να έρθω εδώ και να, και να διαβάσω αυτήν την εξαιρετική μελέτη της ε, κυρίας Ταβέντα. Είναι, πιστεύω, μια ε, πολύ καλή μελέτη που συμπληρώνει όλες τις υπόλοιπες ε, που έχουν γίνει για τον Brexit μέχρι τώρα και ε, ασχολείται και, με, και με, μερικά, με μερικά από τα δικαιώματα των πολιτών. Ε, πρέπει να σας πούμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκτιμά πάρα πολύ ε, την δουλειά σας έτσι ώστε να καταλάβουμε καλύτερα τον Brexit, τις προκλήσεις και τον αντίκτυπο στη ζωή πολλών εκατομμυρίων πολιτών. Εδώ γίνεται λόγος κυρίως για δικαιώματα, όμως νομίζω πως πρέπει να πάμε και πέρα από αυτά και να δούμε πώς επηρεάζει τη ζωή μας, τη δουλειά μας, την ποιότητα ζωής. Πράγματα δηλαδή που δεν σχετίζονται άμεσα με τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών. Και επίσης να σας ασφαλίσω ότι η προστασία των ατομικών δικαιωμάτων είναι κάτι που όλοι εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρούμε θεμελιώδες δικαίωμα για την... Ε, εντάξει, είναι κάτι που πρέπει να ε, διέπει όλες τις ε, διαπραγματεύσεις. Είναι θεμελιώδης αρχή της Ένωσης και να ξέρετε ότι όλοι θα το πάρουμε πάρα πολύ ε, στα σοβαρά. Θα είναι το κύριο μέλημα των διαπραγματευτών. Και οι συνάδελφοι εδώ δεν θα εκπλαγούν όταν τους πω ότι ε, τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών είναι κάτι που δεν ε, συζητήσαμε καν, είναι αυτονόητο. Είναι η ύψιστη προτεραιότητα των διαπραγματεύσεων αποχώρησης του Βασιλείου. Και υπάρχει συνένεση όχι μόνο στο Κοινοβούλιο, αλλά πλήρης συνένεση όλων των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Αυτό είναι κάτι που δεν συμβαίνει συχνά. Έχουμε δείξει την ενότητά μας. Αυτή η ενότητα των 27 κρατών μελών είναι εκπληκτική. Κύριο μέλημά μας είναι τα δικαιώματα των πολιτών λοιπόν γι' αυτό και με χαροποίησε πάρα πολύ που στην μελέτη της καθηγήτριας τα Βέντα αναφέρθηκαν πολλά ζητήματα που σχετίζονται με τις επιπτώσεις και τις συνέπειες του Brexit βασισμένα όμως σε συγκεκριμένα ε, στοιχεία, συγκεκριμένες περιπτώσεις, ε, παραδείγματα. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ε, χρήσιμο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όχι μόνο σε αυτήν εδώ την Επιτροπή, προσπαθούμε ε, να είμαστε ανοιχτοί, να ακούσουμε όσο το δυνατόν περισσότερες φωνές, έτσι ώστε να κατανομήσουμε καλύτερα ε, την κατάσταση και να κερδίσουμε στο τέλος των διαπραγματεύσεων. Ε, ακούμε επίσης πολλούς εμπειρογνώμονες, πολλούς ειδικού ευρωπαϊκού δικαίου. Μας είπαν ότι υπάρχει περιορισμένη νομολογία, δεν υπάρχει προηγούμενο τέτοιο τέτοιου μαζικού αριθμού ανθρώπων ε, που ε, αλλάζει ξαφνικά το καθεστώς του αλλάζει ξαφνικά η ζωή τους από τη μια μέρα στην άλλη. Αυτό είναι μια αναφρηγουμένου περίπτωση που πρέπει να ε, χειριστούμε όχι μόνο από την ανθρώπινη διάσταση αλλά και νομικά. Πολλές φορές η Σεσίλια, η πρόεδρος Επιτροπής Αναφορών, ε, μας ενημερώνει για περιπτώσεις αναφορών που ε, είναι σχετικές με αυτό και βλέπουμε ότι υπάρχει υψηλό επίπεδο ανησυχίας. Ανησυχούμε πάρα πολύ. Ε, γι' αυτό λοιπόν θέλω να σας στείλω ένα μήνυμα και να σας πω πως εμείς θα παλέψουμε για αυτά που έχει καταφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τα δικαιώματα που έχει καταφέρει να δώσει στους πολίτες της. Είναι ε, αναμφισβήτητη και ανεκτήμητη αξία τους. Επίσης, η μελέτη της κυρίας Σταβέντα δείχνει ότι το θέμα αυτό είναι περίπλοκο, ιδιαίτερα ε, εν ώψη των εξελίξεων. Αυτές οι περιπτώσεις ε, με τις οποίες θα ασχοληθείτε είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσες, πολύ σημαντικές. Νομίζω πως ε, πρέπει εμείς ως πολιτικοί να εγγυηθούμε την απόλυτη, τη μέγιστη συνέχεια, να εγγυηθούμε ασφάλεια, σιγουριά στους ε, πολίτες. Γι' αυτό λοιπόν ε, το έγγραφο θέσης το οποίο ε, συστάθηκε από το Κοινοβούλιο και από την Επιτροπή σας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ελπίζουμε λοιπόν να μην διαταραχτεί αυτή η συνέχεια, αυτή η ομαλότητα να μην διαταραχτούν οι διαπραγματεύσεις. Να είστε όμως σίγουροι πως αυτές οι διαπραγματεύσεις θα είναι ε, αποφασιστικής σημασίας. Άρχισαν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην σταματήσουμε την επικοινωνία, να μας ενημερώνετε συνεχώς και πρωτού τελειώσω να σας πω ότι υπάρχουν ε, διαφορετικές στρατηγικές. Έχουμε ακούσει εμπειρογνώμονες, ειδικού ε, εμπλεκόμενους για το τι συμβαίνει. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μια στρατηγική η οποία θα προστατεύσει τα δικαιώματα των πολιτών, ακόμα και αν δεν διατηρούν οι Βρετανοί το ε, την ιδιότητα του πολίτη της Ένωσης προσπαθούμε να ε, διατηρήσουν τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτό και προσπαθούμε επίσης ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να δράσουμε. Έχουμε κατεβάσει ένα ψήφισμα το οποίο ζητά να διατηρηθούν τα δικαιώματα των βερτανών πολιτών. Υπάρχει κάποια σύνδεση ε, με την ε, ιδιότητα του υπηκόου της Ένωσης. Αυτά είναι επιλογές που εξετάζουμε, δεν είναι τίποτα ακόμα σίγουρο. Κυριαρχία, βεβαιότητα, κανείς δεν ξέρει ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Και για να ολοκληρώσω, να πω ότι η εμπειρία σας η συνεισφορά σας με την, τις έρευνες, ε, με όλα όσα κάνετε στην Επιτροπή Αναφορών είναι πολύ σημαντική για τις διαπραγματεύσεις. Αλλά το να σας ακούμε εδώ ζωντανά νομίζω πως ε, βοηθά πάρα πολύ εμάς τους ε, νομοθέτες στο Κοινοβούλιο. Και είναι και ένα δίδαγμα για το πώς εξελίσσεται ε, η έννοια αυτή της ε, ευρωπαϊκής ε, υπηκότητας. Υπάρχουν θέματα στα οποία παρουσιάζουμε ελλείψεις, πρέπει να εφαρμόσουμε τους νόμους, υπάρχουν οι μελλοντικές μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την εμπειρία που θα μας δώσετε εσείς έτσι ώστε να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε την κατάσταση των, της υπηκότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Ντανούτα. Και πάλι βλέπουμε ότι το θέμα του Brexit αφορά ολόκληρο το Κοινοβούλιο, όλες οι επιτροπές και βεβαίως η Επιτροπή ΑΦΚΟ εκεί πέρα θα παίξει τον κύριο ρόλο, αλλά όλοι, όλες οι επιτροπές έχουν εξίσου μεγάλη σημασία έτσι ώστε να υπάρχει δημοκρατικός έλεγχος σε όλη την διαδικασία. Σας ευχαριστώ λοιπόν και πάλι Ντανούτα. Υπάρχουν συνάδελφοι που έχουν ζητήσει τον λόγο, αλλά θα ήθελα αυτή τη στιγμή να περάσουμε στους αναφέροντες για να διευρύνουμε λίγο την συζήτηση. Λοιπόν, έχουμε πρώτα απ' όλα τον αντίκτυπο του δημοψηφίσματος στην ευρωπαϊκή υπηκότητα και στους ευρωπαίους υπηκόους που κατοικούν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Έχουμε πρώτα απ' όλα την αναφορά 0923 του τη Κορίν Μπάιρον Ντανούσερ σχετικά με διατήρηση δικαιωμάτων ε, πολιτών που μένουν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν είναι παρούσα, αλλά ανησυχεί για το ότι τα άτομα τα οποία έδρασαν καλή την πίστη, όπως επεσήμανε η κυρία Σπαβέντα, επηρεάζονται πολύ από το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος και λέει ότι πρέπει να υπάρχει μια εγγύηση των δικαιωμάτων και όχι αναδρομική αφαίρεσή τους. Όλες οι σημερινές αναφορές θα παραμείνουν ανοιχτές για προφανείς ε, λόγους. Η επόμενη λοιπόν είναι η 14-19 του κυρίου Παϊκόπουλου για το ίδιο ακριβώς ε, ζήτημα. Δεν είναι εδώ παρόν ε, και αυτός ανησυχεί πάρα πολύ για το ίδιο ακριβώς πράγμα. Αυτός όμως ε, έχει ε, ασφάλεια υγείας ε, και το δικαίωμα να ψηφίσει, οπότε θεωρεί ότι δεν μπορούν να του αφαιρεθούν τα δικαιώματα που έχει ως πολίτης, καθώς αυτό θα του αφαιρέσει και τα δικαιώματα που προκύπτουν από την ευρωπαϊκή ηθαγένεια. Μετά έχουμε τον κύριο Γνάσιο Ρομέρο Ρομέρο, η αναφορά 470 με 6.139 υπογραφές για την εγγύηση των δικαιωμάτων στο Ηνωμένο Βασίλειο και των Βρετανών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι εδώ ο κύριος Ρομέρο Ρομέρο. Θα έχετε λοιπόν τρία λεπτά εσείς και τρία λεπτά ο κύριος Μπιλάλ Σαμπίρ. Σας ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα, σας ευχαριστώ που μας επιτρέπετε να παρουσιάσουμε την αναφορά μας, μια αναφορά η οποία αρχικά είχε υποβληθεί ε, στο wemove.eu και έχει ήδη συλλέξει 6.000 υπογραφές. Ξεκινήσαμε λοιπόν μια οργάνωση Εσπανιόλες Ερενεωνίδο, Ισπανών στο Ηνωμένο Βασίλειο και ταυτόχρονα μια ομάδα Βρετανών στην Ισπανία, αλλά νομίζω ότι το θέμα της αναφοράς μας αφορά όλους τους ε, Ευρωπαίους πολίτες του και τους Βρετανούς στις 27 άλλες χώρες. Λοιπόν, ας περιγράψω πώς έχει η κατάσταση. Όπως ξέρετε, από το δημοψήφισμα πριν από ένα χρόνο ακριβώς, πολλοί μετανάστες, πολίτες της Ένωσης ε, αγωνιούν ε, γιατί δεν υπάρχουν εγγυήσει για το καθεστώς διαμονής μας στις χώρες που έχουμε μετικήσει. Παρά λοιπόν το ότι δεν απαιτείται από το Ηνωμένο Βασίλειο, πολλοί πολίτες του ΕΟΧ αποφάσισαν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους ζητώντας μία άδεια παραμονής ή ε, κάρτα παραμονής. Όμως ε, υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό των ατόμων αυτών των αιτήσεων που απορρίπτονται αυτή τη στιγμή από το Υπουργείο Εσωτερικών και δεν υπάρχει κάποια εγγύηση αναγνώρισης του καθεστώτος αυτού όταν θα ε, έχουμε τελικά το Brexit επιπλέον. Μεγάλο τμήμα των κοινοτήτων μας δεν μπορεί να εκπληρώσει τις απαιτήσει της ασφάλισης υγείας που είναι αναγκαία για να έχει κάποιος ε, άδεια παραμονής. Τα άτομα αυτά περιλαμβάνουν φοιτητέ, ε, γονείς, ε, άτομα που φροντίζουν άλλους ε, κλπ. Το Ηνωμένο Βασίλειο δεν έχει εφαρμόσει αυτή την απέτηση ασφάλισης υγείας για τα άτομα τα οποία είναι οικονομικά ανενεργά στο παρελθόν ενώ επιλέγει το ότι το NHS θα συνεχίσει να είναι ανοιχτό για όλα τα άτομα τα οποία κατοικούν στην χώρα. Οπότε οι μετανάστες ε, θα χωριστούν σε δύο κατηγορίες. Αυτοί οι οποίοι είναι νόμιμοι, δηλαδή αυτή τη στιγμή εργάζονται ή πληρούν τις ανάγκες ασφάλισης υγείας και αυτούς οι οποίοι δεν ε, συμμορφώνονται με τις απαιτήσει. Και πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη στις διαπραγματεύσεις ε, για τα δικαιώματα της δεύτερης ομάδας όσοι εγκαταστάθηκαν πρόσφατα στην ε, χώρα κινδυνεύουν περισσότερο όσον αφορά τα δικαιώματα τους. Εάν, υπάρξει, εάν δεν υπάρξει συμφωνία στις διαπραγματεύσεις. Συμφωνούμε εδώ πέρα και συμφωνούμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι η καταληκτική ημερομηνία για τους μετανάστες θα πρέπει να είναι η ημερομηνία εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση. Επίσης, ε, άλλοι μετανάστες έχουν σκεφτεί να ζητήσουν υπηκότητα για να προστατευτούν. Όμως κάποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν δέχονται την διπλή υπηκότητα ή εάν το δέχονται λένε ότι θα πρέπει να είναι σε δύο χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιπλέον σε κάποιες χώρες όπως την Ισπανία τα άτομα τα οποία έχουν λάβει την ε, υπηκότητα πρέπει να αποκηρύξουν την προηγούμενη τους υπηκότητα. Κάτι το οποίο είναι πάρα πολλά άτομα. Όπως είπα λοιπόν, έχουμε θέσει κάποια ζητήματα. Θέλαμε να υπάρξει μια επίσημη εγγυήση προς όλους, προς όλους λέω, οι πολίτε που επηρεάζονται από το Brexit ε, βεβαίως, αλλά και να αποφεύγουμε όρους όπως νόμιμη παρανομή που χωρίζει σε κατηγορίες και να υπάρξει ένα σύστημα βίζας εργασίας για όσους κατοικούν ήδη. Επιπλέον, όχι μόνο για όλους τους πολίτες, αλλά θα πρέπει να ε, διατηρηθούν όλα τα βασικά δικαιώματα για τους μετανάστες όπως η παροχή υγείας ή η συντάξη. Πλέον αναγνωρίζουμε ότι βεβαίως το θέμα της υπηκότητας είναι προνόμιο των κυρίαρχων κρατών θα θέλαμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναγνωρίσει την διπλή υπηκότητα για τον πληθυσμό που επηρεάζεται λόγω της εξαιρετικής περίστασης της αποχώρησης του Ενμούνου Βασιλείου και επιπλέον πέρα από τις ε, διαπραγματεύσεις αυτές ζητάμε οι διαπραγματεύσεις να είναι ανεξάρτητες από τα ζητήματα τα οποία αφορούν οτιδήποτε άλλο όπως το εμπόριο ή άλλα ζητήματα για να μην υπάρχει η δυνατότητα να μην καταλήξουμε σε συμφωνία για τα δικαιώματα των πολιτών. Οπότε πρώτα οι πολίτες, αλλά και κυρίως οι πολίτες. Σας ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Ξέχασα, λέει η Πρόεδρος, ότι έχουμε άλλο έναν αναφέροντα, ο κύριος Μπιλάρ Σαβίρ. Παρακαλώ έχετε το λόγο να συμπληρώσετε. εκπροσωπώ μια ομάδα του Αυγούστου 16 μετά από το Brexit. Προσφέρουμε υποστήριξη σε γύρω 20.000 ε, πολίτες ήταν μακριά του μικρόφωνο του κυρίου. Το Ενωμένο Βασίλειο φιλοξενεί περίπου 3,5 εκατομμύρια Ευρωπαίους πολίτες. Είναι πολύ ενισχυτικό ότι ένα χρόνο μετά το δημοψήφισμα αυτοί οι πολίτες της Ένωσης ακόμα δεν γνωρίζουν τι θα γίνει με την κατάστασή του. Και υπάρχουν ευάλωτε ομάδε που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Καταρχάς, οι πολίτε Ένωση που δεν έχουν δικαίωμα, που δεν έχουν διαμονή αλλά διαμένουν και μετά οι πολίτες με αναπηρία και αυτοί που είναι ανασφάλιστοι. Μετά και τα μέλη των οικογενειών αυτών των ανθρώπων. Στον Ηνωμένο Βασίλειο η κυβέρνηση έχει εφαρμόσει νομοθεσία που μεταφέρει τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Δυστυχώς όμως, όταν αυτά τα άτομα ζητούν άδεια διαμονής, υπάρχει υπερβολική γραφειοκρατία. Το έντυπο, το αντιστοιχό είναι 85 σελίδες και από το Φλεβάρι φέτος θα πρέπει να καταγραφούν το οποίο σημαίνει ότι οποιαδήποτε αίτηση δεν έχει συμπληρωθεί, έστω και να έχει συμπληρωθεί ένα τετράγωνο, σημαίνει ότι υπάρχει ένα τέλος διοικητικό 25 λιρών που επιβάλλεται. Και επίσης δεν λαμβάνεται υπόψη γεγονότα όπως το κατά πόσο έχουν οικογενειακούς δεσμούς με τις χώρες ε, καταγωγής τους. Επίσης, οι ετώντε θα πρέπει να υποβάλουν συνεχώς έγγραφα, κάτι το οποίο είναι προβληματικό, ιδιαίτερα για αυτούς που βασίζονται σε ιστορικά αναλογικά στοιχεία. Το 2008 δεν υπήρχε κανένα διοικητικό τέλος και το έντυπο το αντίστοιχο ήταν 13 σελίδε. Δεν υπάρχουν εξελίξεις νομοθετικέ στην Ένωση που να δικαιολογούν κάτι τέτοιο. Τα τωρινά διοικητικά μέτρα σημαίνουν ότι αποτρέπονται από το να υποβάλουν αίτηση για άδεια διαμονής οι πολίτες της Ένωσης και αυτό βεβαίως αποτελεί μια παράνομη παρέμβαση στην, στο δικαίωμα κυκλοφορία. Θεωρούμε λοιπόν θα πρέπει να βελτιώσουμε το σύστημα. Αν δούμε υπόψη μα την Ιρλανδία ως αντίστοιχη χώρα, βλέπουμε ότι τα έντυπα τα δικά του είναι τις 3,5 σελίδες και ότι δεν εφαρμόζουν τα αποδεικτικά αρχικά στοιχεία, το οποίο σημαίνει ότι μπορούν να λάβουν ε, ταυτότητα στη διαβατήρια κατά τη διάρκεια όλη τη διαδικασία. Δεν υπάρχει λοιπόν λόγο για να μην θετήσει παρόμοια προσέγγιση η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου. Το 2011 επίση το Ηνωμένο Βασίλειο επέβαλε την υποχρέωση για α, ιατρική περίθαλψη στους πολίτες της Ένωσης. Παρ' όλα αυτά αρνήθηκε να προσφέρει πρόσβαση σε πολίτε ένωσης, σε πολίτες Βρετανούς εκτός Βρετανίας. Και γι' αυτό ακριβώς ξεκίνησε μια διαδικασία παράβαση κατά του Ηνωμένου Βασιλείου, που έβρισκε σε εξέλιξη. Επίσης, όταν απαιτείται αυτή η ιατρική περιθέλψη, για αυτούς που δεν τη διαθέταν, βρισκόταν σε μια κατάσταση αδυναμίας και δεν μπορούσαν να φροντίσουν σε αυτούς τους. Αυτό περιλαμβάνει οποιοδήποτε πολίτη τη Ένωσης που διέμενε στο Ηνωμένο Βασίλειο επί δεκαετίες και που, ήταν, και που είχαν εισοδήματα. Ακόμα και τις νοσοκόμες αφορά αυτό ή και άλλες κατηγορίες ανθρώπων. Αυτά τα άτομα λοιπόν δεν έχουν δικαίωμα άδειε διαμονή και βρίσκονται σε μια ευάλωτη κατάσταση. Και δεν μπορούν παρά να δαπανίσουν πάρα πολλά χρήματα για να τακτοποιηθούν. Αυτούς ακριβώς θα πρέπει λοιπόν να καλύπτει και να προβλέπει το, η νέα νομοθεσία. Αναμένω λοιπόν το αποτέλεσμα αυτό των διαπραγματεύσεων αυτές τις κατηγορίες ανθρώπων ώστε να δοθούν ε, εγγύσει και να διασφαλιστούν αυτοί οι άνθρωποι. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα θα αρχίσουμε τη συζήτηση. Όπως είδατε όμως, Σας παρακαλώ να είστε πολύ ακριβείς στις παρεμβάσεις σας και στις ερωτήσεις σας. Ε, θα πρέπει να τελειώσουμε στις 12.30 ε, και έχουμε αρκετές αναφορές. Οι 11, αφορούν το ίδιο θέμα. Θα παραμείνουν ανοιχτέ. Λείπουν βεβαίω οι αναφέροντε. Αλλά θα δώσω λόγο καταρχά στην κυρία Άντερσον και στην κυρία Σπινέλη από την Επιτροπή μα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για την ε, ευκαιρία που μου δίνετε να σας μιλήσω σήμερα. Είμαι ευρωβουλευτής από τη Βόρεια Ιρλανδία και θα ήθελα να σας μιλήσω σε σχέση με το τμήμα 6, αυτό που ονομάζουμε Ιρλανδικές ιδιαιτερότητες. Αλλά αυτό εντάξει είναι και το καινούργιο. Με ενδιαφέρει ιδιαίτερα το 3-5 άρθρο και το άρθρο 8 ε, της Διεθνούς Συνθήκης που επιτρέπει δηλαδή Ιδιαίτερε συνθήκε με τις γειτονικέ χώρε τα άρθρα 9 και τα άρθρα 10. Εδώ, όταν μιλάμε για το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, αυτό μίλησε για τα δικαιώματα άσκηση ψήφου στις ευρωεκλογέ σε τρίτη χώρα. Για κάποια από τα θέματα που αφορούν την Βόρεια Ιρλανδία νομίζω δεν δίνουν ιδιαίτερη προσοχή. Εγώ το που διαθέτω στο ταξιδικό έγγραφο είναι ένα Ιρλανδικό διαβατήριο και όλοι έχουν στη Βόρεια Ιρλανδία Ιρλανδικό διαβατήριο παρόλο που βρισκόμαστε υπό την δικαιοδοσία της Βρετανίας. Οπότε μετά το Brexit, παρά συμφωνία της ε, Παρασκευής, θα βρεθούμε σε δυσμενή θέση. Οπότε θα πρέπει να δούμε ακριβώς τι γίνεται και τι είναι απαραίτητο να γίνει όσον αφορά την τρόπο στο πρωτοκόλλο. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν τι γίνεται με τα δικαιώματά μας, γιατί ως Ιρλανδός υπηκός με ευρωπαϊκό διαβατήριο και με ευρωπαϊκά δικαιώματα, θέλω να είμαι βέβαιος ότι το 1,8 εκατομμυρίων πολιτών στη Βόρεια Ιρλανδία θα καλυφθούν σε αυτή τη φάση διαπραγμάτευσης και δεν θα παρακαμφθούν ή δεν θα ξεχαστούν και θα μείνουν στο πλαίσιο των Ιρλανδικών ιδιαιτεροτήτων. Ευχαριστώ κυρία Σπινέλη. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Ευχαριστώ την συγκήτρια, την καθηγήτρια Σπαβέντα. Ευχαριστώ και τους εκπροσώπους των αναφορών που αποδεικνύονται ένα ουσιαστικό στοιχείο κατά τη διάρκεια αυτής της διαπραγμάτευσης. Μια ερώτηση θα ήθελα να κάνω στην κυρία Σπαβέντα. Νομίζω ότι θα πρέπει να προβλέψουμε διάφορες δυνατότητες όσον αφορά τους χρονισμούς και να μην αποκλείσουμε την, το ενδεχόμενο βραχυπρόθεσμα να μην πετύχουμε συμφωνία. Ιδιαίτερα εάν πέρα από τις εκλογές που είχαμε, αν θα έχουμε μάλιστα και σε εξπερικούς χρόνους λύσεις διαφορών στο εσωτερικό των συντηρητικών Φαντάζομαι λοιπόν ότι θα χρειαστεί μια μεταβατική συμφωνία για να αποφύγουμε ακριβώς αυτό το κενό. Σε αυτή λοιπόν τη μεταβατική περίοδο θα ήθελα να ρωτήσω πώς θα εφαρμοστεί η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία θα ισχύει και κατά διάρκεια μεταβατική συμφωνίας και θα πρέπει να δώσουμε μάχη επ' αυτού και εδώ περιλαμβάνω και το βασικό για μένα δηλαδή τον έλεγχο του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που ασκείται δηλαδή από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ακριβώς για να προστατεύσουμε όλα τα δικαιώματα όλα αυτά τα δικαιώματα που διατρέχουν τον κίνδυνο να εξαφανιστούν αν η μεταβατική συμφωνία δεν κυριαρχείται από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και από το Δικαστήριο. Αν δεν ισχύσει δηλαδή όλη η προϋπάρχουσα νομολογία του Δικαστηρίου με ενδιαφέρει επίσης πάρα πολύ αυτό που είπατε για τον ορισμό των εργαζομένων που από ό,τι κατάλαβα στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία ο ορισμός είναι πολύ προχωρημένος και θα ήθελα να καταλάβω αν αντίστροφα βρίσκεται στην τελείως διαφορετική θέση στο Ρωμαίο Βασίλειο. Και κάτι άλλο τελευταίο. Βλέπω ότι η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσει μια διαδικασία καταγραφής των Ευρωπαίων πολιτών. Τρία εκατομμύρια περίπου είναι αυτή Θα ήθελα να μάθω αν πράγματι υπάρχει κάποιο πρόβλημα μη συσχετισμού αυτής της διαδικασίας καταγραφής με το δικαίωμα διαμονής μόνιμης διαμονής στη χώρα. Γιατί από ό,τι κατάλαβα, αυτή η διαδικασία καταγραφής, επειδή ακριβώς δεν παρέχει επαρκείς εγγυήσεις για την διαμονή, οθεί πολλούς Ευρωπαίους πολίτες να μην καταγραφούν, να αρνηθούν την καταγραφή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριο Σπρέντα. Ευχαριστώ πολύ. Δυστυχώς δεν έχουμε πολύ χρόνο και θα πρέπει να φύγω. Εγώ θα ήθελα να αναφερθώ στην, στην αναφορά που μας παρουσίασαν οι δύο αναφέροντες και που αφορά το καθεστώς των Ευρωπαίων πολιτών στην Μεγάλη Βρετανία, όπως είπε και η Πρόεδρος. Δεν θα αναφερθώ σε λεπτομέρειε των αναφορών, θα κάνω μια πρόταση. Δηλαδή, το Κοινοβούλιο να προετοιμάσει ένα ψήφισμα το οποίο θα επικεντρώνεται στα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών που διαμένουν στην, στην Μεγάλη Βρετανία. Συγγνώμη. Θα πρέπει λοιπόν να επικεντρωθούμε ως Κοινοβούλιο στον σεβασμό των θεμελιωδών ελευθεριών των πολιτών της Ένωσης που βρίσκονται στη Μεγάλη Βρετανία και που κινδυνεύουν από το 19 και μετά. Προτείνω λοιπόν, προτείνω λοιπόν να κάνουμε αυτό το ψήφισμα. Και συγγνώμη που πρέπει να φύγω. Ωραία. Αυτό το ψήφισμα προβλέπεται για μετά τις θερινές διακοπές. Ε, κυρία Τάρλινγκ. Ε, ε, ευχαριστώ. Έχω και εγώ μερικά θέματα, μερικά σχόλια. Θα τα κάνω έτσι ανα θέμα. Αρχίζω λοιπόν. Η Ντανούτα είπε κάτι πάρα πολύ σημαντικό, διότι πολύ συχνά μιλάμε για τα δικαιώματα ε, των ε, πολιτών της Ένωσης, αλλά μιλάμε για ανθρώπινες ζωές, μιλάμε για ανθρώπους. Πολλοί επηρεάζονται με πολλούς ε, τρόπους. Εμείς εδώ οι Βρετανοί που μένουμε στο Βέλγιο, δεν ξέρουμε ποιο θα είναι το μέλλον μας, δεν ξέρουμε τι ε, μας επιφυλάσσει το μέλλον. Ε, και είναι πολλοί σαν και εμάς, οι οποίοι χρησιμοποίησαν το δικαίωμα του πολίτη της Ένωσης. Προσπάθησαν να το ε, χρησιμοποιήσουν στο ΕΡΕΠΑΚΡΟΝ και τώρα είναι λες και μας τράβηξαν το χαλί κατά τα πόδια. Ε, είμαστε στον αέρα. Και πρέπει να πω ότι είναι ντροπή ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν έλαβε κάποια απόφαση αμέσως μετά το δημοψήφισμα έτσι ώστε μονομερός έστω να δώσει κάποια ε, διασφάλιση στους πολίτες ε, της, να ξέρει ποιο είναι το μέλλον τους και περιμένει μέχρι τώρα, μέχρι τις διαπραγματεύσεις και αυτή είναι και η προσωπική μου θέση ως ε, Βρετανίδα Ευρωβουλευτής αλλά ε, πραγματικά θεωρώ πως είναι λυπηρό που δεν υιοθετήθηκε στο μία μονομερή σε απάντηση άσχετα με αυτό που θα γίνει. Τώρα, δύο σημεία να πω ότι ω Επιτροπή Αναφορών πρέπει να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε με τι αναφορέ. Και εγώ θα ήθελα να δω ε, τα εξή. Η μελέτη τη ε, καθηγήτρια Παβέντα είναι εκπληκτική. Αυτό που ακούσαμε σήμερα το πρωί ήταν ε, τόσο εκπληκτικό όσο και τρομακτικό πραγματικά είναι μια καυκική ε, κατάσταση. Δεν ξέρουμε τι μας επιφυλάσσει το μέλλον, όλα είναι αβέβαια. Υπάρχει ένα συνονθήλευμα ε, προτάσεων και γι' αυτό λοιπόν εγώ θέλω να πω σε όσους είναι πολιτικά υπεύθυνοι για την έκθεση για τα πολιτικά δικαιώματα των πολιτών, κυρία Χούμπνερ εσείς θα είστε στο επίκεντρο αυτής της έκθεσης, να σας πω ότι θα υπάρχουν άτομα από κάθε πολιτικές ομάδες, αλλά οι πληροφορίες πρέπει να φτάνουν στα χέρια των ευρωβουλευτών, έτσι ώστε να διασφαλίσουμε ότι η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα είναι το όσο, όσο το δυνατόν ευρύτερη, θα καλύπτει όσο το δυνατόν περισσότερου τομείς. Τώρα, κάτι διαδικαστικό αλλά εξίσου σημαντικό. Νομίζω πω πρέπει να στείλουμε μια επιστολή στην κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου που θα τονίζει τι λεπτομέρειε που αντιμετωπίζουν οι Βρετανοί πολίτε τώρα σε ό,τι αφορά την ε, διαμονή τους και τα δικαιώματά τους. Είναι πολύ σημαντικό να διατηρήσουμε το ρόλο μας ε, ως Επιτροπή Αναφορών, ε, να πάρουμε τους εαυτούς μας στα σοβαρά και να μεταφέρουμε αυτό το μήνυμα των αναφερόντων στην κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου. Τώρα, παράλληλα με τις διαπραγματεύσεις. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να προτείνω αυτές τις δύο δράσεις και ελπίζω να μιλώ και εκ μέρου των συναδέλφων μου, αλλά εκ μέρου των ε, Βρετανών Ευρωβουλευτών θα ήθελα να πω στου αναφέροντε ότι λυπάμαι πραγματικά που έχετε βρεθεί σε αυτή τη θέση. Είναι άδικο και δεν θα έπρεπε να έχει γίνει με αυτόν τον τρόπο. Ε, ευχαριστώ πολύ Τζούντι. Ναι, δεν συμβαίνει συχνά, αλλά σήμερα σε χειροκροτούν ε, οι συνάδελφοι του ΕΛΚ. Να πείστε αυτό. Κυρία Μπεσέρα έχει το λόγο. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ και του αναφέροντε που ήρθαν και που έχω την τύχη να γνωρίζω εδώ και καιρό. Έχουμε συνεργαστεί και στον κυβερνοχώρο και μετά διαζώσεις. Αυτή η 3 εκατομμύρια είναι μια θαυμάσια οργάνωση. Ένα υπόδειγμα θα έλεγα. Έγινε το Brexit, χωρίς να το καταλάβουμε, με τρόπο που δυστυχώς δεν αλλάζει και προκαλεί πολλούς φόβους και αβεβαιότητες. Έχει περάσει ένας χρόνος από το Brexit, από την απόφαση και έχουμε την έκθεση για την ηθαγένεια που κάνουμε κάθε τρία χρόνια και για την οποία είμαι συγγήτρια και σας διαβεβαιώνω ότι θα έχει πολύ σημαντικό χώρο το θέμα του Brexit εκεί. Πέρα πάντως από την απώλεια εμπιστοσύνης αυτών που ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο και των Βρετανών και των πολιτών της Ένωσης, βλέπουμε ότι έχασαν την εμπιστοσύνη στην κυβέρνησή τους. Έφτασαν σε καταστάσεις απελπισίας για τη διασφάλιση της ε, διαμονής τους και θα δούμε πώς θα εξελιχθούν εκεί τα πράγματα. Και νομίζω ότι η σχέση εμπιστοσύνη που ε, είχαμε με τα θεσμικά όργανα ήταν πολύ σημαντική. Νομίζω ότι με την αρχική όθηση του Κοινοβουλίου καταφέραμε να δημιουργήσουμε μια εμπιστοσύνη που επικυρώθηκε από το Συμβούλιο και την Κομισιόν και με το διαπραγματευτή μας. Το Citizens First, το πρώτο οι δεν είναι απλό σλόγγ, αλλά είναι μια πεποίθηση που θα προσπαθήσουμε να εφαρμόσουμε και να επενθυμίσω ότι εμείς ως Επιτροπή Αναφορών έχουμε δεσμευτεί να κάνουμε άλλη μια ακρόαση το καλοκαίρι σε συνδυασμό με άλλες επιτροπές και νομίζω ότι η, διαπραγματε... η διαπραγμάτευση ακριβώς θα είναι κεφαλαιόδου σημασία όσον αφορά την ασφάλιση των δικαιωμάτων. Και χαίρομαι που πρόσφατα είχαμε μεγάλο αριθμό πολιτικών ηγετών που θεωρούν ότι είναι αναστρέψιμο το Brexit. Ο ίδιος ο συντάκτης του άρθρου 50 το είπε πρόσφατα και είπε ότι αν αλλάξουμε τον τρόπο σκέψης για την αποχώρηση μπορούμε να το κάνουμε και κανείς ε, στις Βρυξές δεν μπορεί να μας σταματήσει. Αυτό λοιπόν το οποίο φαινόταν ε, γραμμένο πάνω σε... στην πέτρα πρόσφατα από τις Βρυξέλλες είπαν ότι αν θέλετε να κάνετε μια υποχώρηση τότε, εντάξει, πολύ ωραία, Εμεί είμαστε εδώ για να δημιουργήσουμε μια ισχυρή Ευρώπη. Όντω μπράβο στου πολίτε οι οποίοι πραγματικά κάνουν καθημερινά μεγάλε μάχε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Μπέτρη. Τώρα να δώσω τον λόγο στην κυρία Σκότ κάτω εξ μια μια διαφορετική επιτροπή για το ίδιο θέμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε που μου δίνετε τον λόγο. Χτες ήμουν σε μια παρουσίαση κάποιων δικηγόρων από το Πανεπιστήμιο του Σουάντσι εξ για μια έκθεση που είχαν αναθέσει οι πράσινοι για τους G11 ε, και αφορά ακριβώς ε, τα δικαιώματα των δύο αυτών κατηγοριών πολιτών ε, στην, σύμφωνα με την σύμβαση της Βιέννης. Είχα ακούσει ε, διάφορα πράγματα κατά τη διάρκεια του δημοψηφίσματος. Λοιπόν, υπάρχει αυτή η μελέτη από τον Τζιλ Evans και λένε ότι αν έχεις ε, γεννηθεί πριν φύγουμε από την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση, όλοι έχουν αυτά τα δικαιώματα. Σας ευχαριστώ. Ναι, θα το εξετάσουμε και θα ήθελα να μας δώσετε πληροφορίες γραπτός. Θα βοηθήσει νομίζω την γραμματεία. Μάλιστα, σας ευχαριστώ κύριος Γιάρ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα εγώ τουλάχιστον η σημερινή συνεδρίαση να μεταδίδεται απευθεία στην Βρετανική κυβέρνηση. Από ό,τι φαίνεται ότι, φαίνεται ότι δεν θα υπάρχουν κερδισμένοι από το Brexit. Αυτό διαπιστώνουμε. Και προσπαθούμε τώρα να περιορίσουμε τις ζημιές. Και ε, έχουμε... Μιλήσαμε για όλα αυτά τα πράγματα. Έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε. Οι οικονομικές σχέσεις, ε, διεθνείς σχέσεις εσωτερική πολιτική, αλλά δεν θα πρέπει πράγματι τα δικαιώματα των πολιτών να αποτελέσουν ένα διαπραγματευτικό χαρτί. Χρειάζεται να υπάρχει κάποια εμπιστοσύνη, γιατί τα προβλήματα τα οποία έχουμε εμφανίστηκαν ε, γιατί ακριβώς αυτοί οι άνθρωποι πίστεψαν στην σκέψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν επιτρέπεται να τους να καταστρέψουμε αυτή την εμπιστοσύνη. Όπως είπατε, τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν μπορεί να μπαίνουν στο ζύγι της διαπραγματευσής. Έχουμε ήδη αρκετά προβλήματα. Ε, πρέπει να ληφθούν αυτά υπόψη από την Βρετανική κυβέρνηση και εμένα με ενοχλεί λίγο ότι ε, έχω την εντύπωση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ανισχύει περισσότερο από τη Βρετανική κυβέρνηση, ε, επισήμως τουλάχιστον. Ένα ερώτημα προς την ε, κυρία Σπαβέντα. Το ανακοινώσατε αλλά δεν το είπατε γιατί δεν έφτανε ο χρόνος την ειδική σχέση μεταξύ Ιρλανδίας ε, και Βρετανίας με την Βόρεια Ιρλανδία. Γιατί για μένα το πρόβλημα ε, αφορά και την συμφωνία αλλά η Ιρλανδία είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι γίνεται, δεν ξέρω, θα υπάρξει κάποια ειδική οικονομική ζώνη, πώς θα μπορούσαμε να το πούμε. Σας ευχαριστώ. Θα δώσω τώρα τον λόγο ξανά στην ε, κύρια Σπαβέντα για να απαντήσει σε κάποιες ερωτήσεις. Ε, μετά θα ακούσουμε την επόμενη αναφορά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τις ερωτήσεις για το Ιρλανδικό ζήτημα που ρώτησε και ένας άλλος βουλευτής. Ε, είναι ενισχυτική η κατάσταση στην Ιρλανδία για όσους ζουν στη Βόρεια Ιρλανδία και στη Δημοκρατία της Ιρλανδίας. Μέχρι προσφάτως. Τώρα, το τι θα γίνει με τις βίζες. Η Δημοκρατία της Ιρλανδίας δεν είναι στην συνθήκη Σέγγεν, οπότε μπορούν να κάνουν τις δικές τους διευθετήσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο. Και αυτή τη στιγμή περιοχή ταξιδιών μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Δημοκρατίας της Ιρλανδίας προστατεύεται από ένα πρωτόκολλο. Αυτό μπορεί να συνεχίσει και νομίζω πως υπάρχει η πολιτική βούληση για να συνεχίσει να ισχύει. Το πραγματικό πρόβλημα σε σχέση με την Ιρλανδία και τη Βόρεια Ιρλανδία είναι εν μέρη το ζήτημα των Ιρλανδών πολιτών στη Βόρεια Ιρλανδία αλλά και προστασία που παρέχει αυτή τη στιγμή η δημοκρατία της Ιρλανδίας στους Βρετανούς πολίτες και αντιστρόφως που είναι πιο εκτεταμένη από αυτήν η οποία παρέχεται στους ε, Ευρωπαίους πολίτες. Και αυτό μπορεί να είναι πρόβλημα, είναι ήδη πρόβλημα σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, αλλά όταν βγει το Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχει ο κίνδυνος κάποιος να φέρει αυτή την υπόθεση στα δικαστήρια για τη μεταχείριση των Βρετανών στην Ιρλανδία. Οπότε αυτό το οποίο ελπίζω είναι η συμφωνία που θα διαπραγματευτεί το Ηνωμένο Βασίλειο με την Ιρλανδία να αποκτήσει κάθεστος ε, στην ε, συνθήκη, ένα πρωτόκολλο ή να μπει και στην ε, συμφωνία απόσυρσης. Λοιπόν, τώρα η κυρία Σπινέλη είχε ρωτήσει κάτι για το τι θα συμβεί αν δεν, αν δεν καταφέρουμε στα δύο χρόνια να διαπραγματευτούμε και τι γίνεται με τη μεταβατική συμφωνία. Εδώ θα πρέπει να υπάρξει καλή θέληση από το Ηνωμένο Βασίλειο επειδή η μεταβατική συμφωνία θα υλοποιηθεί μόνο αν το επιθυμεί το Ηνωμένο Βασίλειο. Αν αυτοί λοιπόν αποφασίσουν και ειλικρινά νομίζω και εγώ και η πλειοψηφία ημών ελπίζουμε να μην συμβεί, αλλά αν αποφασίσουν να φτάσουμε στο κενό, τότε θα πρέπει να υπάρξει αδιάμεση συμφωνία. Και η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου δεν θα ισχύει πια για το Ηνωμένο Βασίλειο από τη στιγμή που θα φύγουν. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι τα δικαστήρια του Ηνωμένου Βασιλείου δεν θα θελήσουν να προστατεύσουν τους πολίτες. Γιατί η Ευρωπαϊκή Συνθήκη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων θα συνεχίσει να ισχύει και δεν αποκλείεται τα εθνικά δικαστήρια να προσφύγουν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ακριβώς για να ερμηνεύσουν την ε, νομοθεσία μέχρι τη στιγμή που άρχισαν να συμβαίνουν όλα αυτά. Οπότε μετά το Brexit επειδή θα ισχύει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, θα πρέπει τα εθνικά δικαστήρια να κάνουν την ερμηνεία. Πάντως το αγγλικό δικαστικό σύστημα, το οποίο είναι θαυμάσιο, νομίζω θα πράξει σωστά. Το θέμα των εργαζομένων είναι τεράστιο πάντω. Ο ορισμό του εργαζόμενου στο Ηνωμένο Βασίλειο αυτή τη στιγμή ε, συνοδεύεται από αυτέ τι ε, προποθεσει νομιζω Νομίζω 20-30 ώρε τη εβδομάδα εργασία κάτι τέτοιο θυμάμαι λίγο μιλήτρια. Και κάποια ελάχιστα εισοδήματα, ελάχιστε απολαυέ. Στην δική μα την έκθεση, με τη συγκριτική μελέτη όλων των χωρών της Ένωσης πάνω από το ίμιση δεν τηρούσαν την ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Το οποίο σημαίνει ότι όταν θα έχουμε συμφωνία, ελπίζουμε να έχουμε συμφωνία μεταξύ ΙΤΑΒΙΤΑΕ, είναι απαραίτητο όχι μόνο το Ηνωμένο Βασίλειο να αποδεχτεί την ενσωμάτωση του ορισμού του εργαζόμενου, αλλά και όλες οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες να το κάνουν, ας πούμε η Ιταλία, η Σουηδία, ή οποιοδήποτε άλλος. Όχι μόνο το ενωμένο Βασίλειο δηλαδή. Τώρα, για την γραφειοκρατία. Μπορεί να ζητήσει την καταγραφή του Ηνωμένου Βασίλειου και ίσως βρεθούμε σε μια παράδοξη κατάσταση όπου οι πιο γραφειοκρατικές χώρες θα έχουν περισσότερες δυνατότητες να παράσχουν την άδεια αυτή διαμονής από ότι το ενό λοιπόν που τώρα δεν έκανε καταγραφή. Για τα υπόλοιπα, νομίζω κάποιο ανέφερε την εφαρμογή των δικαιωμάτων τη χάρτα και των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Νομίζω ότι αυτό απασχολεί πολλούς από εμά και δεν είναι πολύ τόσο σαφές το τι θα γίνει. Νομίζω ότι ξέρετε, η πρόταση μιας επιστολής ε, προς τον Ηνωμένο Βασίλη για τα διαδικαστικά που έκανε η Α, είναι καλοδεχούμενη γιατί πολλοί νομικοί θεωρούν και εγώ ότι η τωρινή εφαρμογή του καθιστώτος μόνιμης παράνομης δεν ε, συνάδει με το ευρωπαϊκό δίκαιο και ο χρόνος τρέχει και δεν θα μπορέσει να εκδικαστεί μια υπόθεση στο ΔΕΚ για να σταματήσει αυτή την γραφειοκρατική αντιμετώπιση. Αλλά με όλους τους συναδέλφου που μίλησα ούτε ένα δεν θεωρεί ότι αυτή η εφαρμογή συμφωνεί με την οδηγία Οπότε μπορείτε να ρωτήσετε την νομική υπηρεσία, δεν ξέρω, να κοινοποιήσει κάτι. Σας ευχαριστώ και για αυτήν την πληροφορία που θα εκμεταλλευτούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Σπαβέντα, τώρα νομίζω πως ε, μπορούμε να περάσουμε στο δεύτερο τμήμα το οποίο αφορά το μέλλον των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου. Και θα ήθελα να τονίσω ότι Έχουμε την αναφορά 843 του Derek Etherington ε, και την αναφορά 528 ενό Βρετανού πολίτη με τα αρχικά HM. Δεν είναι παρόντες. Το ίδιο και με την αναφορά του 844 του Duncan Parker ο οποίος επίσης απουσιάζει. Για να δούμε τώρα. Επόμενη. Η 803 του LM, επίσης βρετανοητικό δεν είναι ε, ούτε αυτός παρόν. Έχουμε δύο παρόντες που συμφώνησαν να μιλήσουν το απόγευμα. Έχουμε την 790 του Edward Williamson και την 1142 του κυρίου Κάθριτς και συμφωνήστε και οι δύο να μιλήσετε μετά το διάλειμμα για να έχετε αρκετό χρόνο. Και προσέλευση των συναδέλφων βεβαίω που από ό,τι φαίνεται ήδη έφυγαν. Λοιπόν, αυτό θα κάνουμε. Item 24, which is petition 307 by Fiona. Το σημείο 24, η αναφορά 307 της Fiona Godfrey για τα δικαιώματα των Βρετανών πολιτών στις 27 χώρες ε, και των πολιτών των 27 χώρων στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η Jane Golding, ε, πρόεδρος των Βρετανών στην Ευρώπη βρίσκεται εδώ και εκπροσωπεί την αναφέρουσα. Λοιπόν, εάν θέλετε να πάρετε τον λόγο, ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ που μας δίνετε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε την αναφορά μας σήμερα στην Επιτροπή σας. Ε, εξ ε, της Ένωσης Διαφόρων Ομάδων Βρετανών Πολιτών στην Ευρώπη. Να ευχαριστήσω και την καθηγήτρια την κυρία Σπαβέντα για την εξαιρετική παρουσίαση της, ε, της ε, πολυπλοκότητας του θέματος. Η οργάνωση British in Europe είναι μια ένωση 11 οργανώσεων πολιτών με 30.000 ενεργά μέλη στις 27 χώρες. Συνεργαζόμαστε στενά με τις ομάδες των τριών εκατομμυρίων Ευρωπαίων πολιτών στο Ηνωμένο για να διασφαλίσουμε τα δικαιώματα μεταξύ 4 και 5 εκατομμυρίων πολιτών ε, και στις δύο πλευρές ε, της ε, μάχης. Σκοπεύουμε να μην επηρεαστούν αναδρομικά και αρνητικά τα άτομα όταν φύγει το Ηνωμένο Βασίλειο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή είναι η βασική μας αρχή. Όλοι αυτοί οι πολίτες ε, πήγαν σε μια άλλη χώρα καλή την πίστη βασιζόμενοι στα δικαιώματα που είχαν ε, ως ε, Ευρωπαίοι πολίτες. Όλοι είχαν θεμητές προσδοκίες ότι τα συνέχισαν να έχουν αυτά τα δικαιώματα ως πολίτες της Ένωσης για το υπόλοιπο της ζωής τους. Το θέμα λοιπόν είναι θέμα θεμελιώδους δικαιοσύνης και για τις δύο ομάδες. Επιπλέον βρίσκονται σε πολύ δύσκολη θέση ως αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ε, του Brexit και το ότι δεν έχουν ξεκαθαρίσει τα δικαιώματα τους. Εδώ και ένα χρόνο αντιμετωπίζουν μεγάλη αβεβαιότητα, δεν μπορούν να λάβουν αποφάσεις για την προσωπική και την οικογενειακή και επαγγελματική ζωή τους. Βρίσκονται σε ένα κενό, ειδικά οι πιο ευάλωτοι όπως σύνταξη συνταξιούχοι, ε, πλέον έχουν ζητήματα υγείας και πρέπει να το θυμόμαστε αυτό ότι η συντριπτική πλειοψηφία αυτών των πολιτών δεν μπόρεσαν να ψηφίσουν στο δημοψήφισμα παρά το ότι τους επηρεάζει άμεσα. Άρα θα πρέπει να συνεχίσουν ε, οι πολίτες να έχουν τα δικαιώματα που είχαν οι θα είχαν ε, εάν ήταν το Ηνωμένο Βασίλειο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το δικαίωμα παραμονής δεν αρκεί. Τα δικαιώματα που έχουν ως Ευρωπαίοι πολίτες είναι αδιέρετα και τα χρειάζονται όλα για να παραμείνουν στην χώρα όπου βρίσκονται. Με άλλα λόγια, αυτό σημαίνει όλα τα δικαιώματα, όπως το δικαίωμα εργασίας, ε, είτε μιλάμε για εξαρτημένη εργασία ή μη ή την αγνώριση προσόντων ή μεταχείριση το δικαίωμα μετακίνησης μεταξύ όλων των ε, χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς να χάσουν κάποια δικαίωματα δικαίωμα στην ε, ασφάλιση υγείας συντάξεις, κοινωνικές παροχές, ε, το να ψηφίζουν σε ευρωεκλογές και να λαμβάνουν υπηκότητα. Το δικαίωμα να παραμείνουν, παραδείγματος χάρη, δεν ωφελεί έναν επαγγελματία εάν ε, τα επαγγελματικά προσόντα τα οποία χρειάζεται για να ε, εργαστεί πλέον δεν αναγνωρίζονται μετά το Brexit ή εάν δεν μπορεί πλέον να ε, συνεχίσει να έχει την επιχείρησή του. Το ίδιο ισχύει και για τους συνταξιούχους. Το δικαίωμα παραμονής δεν έχει πολύ νόημα για κάποιον ο οποίος δεν δικαιούται πλέον πρόσβαση στο σύστημα δημόσιας υγείας. Ειδικά όταν βρίσκεται σε μια ηλικία όπου η προϋπάρχουσα ασθένεια καθιστά πολύ ακριβή την ιδρυτική ασφάλιση. Έχουμε ασκήσει πίεση στην Βρετανική κυβέρνηση να μην αφαιρέσει αυτά τα δικαιώματα από τους Ευρωπαίους πολίτες στο Ηνωμένο Βασίλειο όταν φέρει τον σχετικό νόμο και να εγγυηθεί, να προσπαθήσει να εγγυηθεί τα δικαιώματα των Βρετανών πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις διαπραγματεύσεις. Το ίδιο αίτημα καταθέσαμε στην κοινή συνάντηση της δικής μας ομάδας και των Ευρωπαίων στο Ηνωμένο Βασίλειο όταν συναντηθήκαμε με τον ε, κύριο Μπαρνιέ την ημέρα που ενεργοποιήθηκε το άρθρο 50 και μετά με την συνάντησή μας με την ομάδα εργασίας του άρθρου 50. Και είχαμε και τη σχετική ακρόαση τον Μάιο. Έχουμε απευθύνει επίσης κοινέ επιστολές με την ομάδα των 3 εκατομμυρίων σε αρχηγούς κρατών ε, των 27 για να ζητήσουμε εγγυήσεις. Όπως ε, και συναντήκαμε με αξιωματούχους και πολιτικούς στις 27 χώρες. Βρετανοί στην Ευρώπη. Λοιπόν, η οργάνωσή μας ε, καλωσορίζει τις ε, κατευθυντήριες γραμμές ε, του Συμβουλίου που υιοθετήθηκαν στις 27 Απριλίου ως ένα τεράστιο βήμα για την διασφάλιση των περισσότερων δικαιωμάτων που επιθυμούμε, όπως επίσης και τις τελικές διαπραγματευτικές οδηγίες και τις βασικές αρχές για τα δικαιώματα των πολιτών, όπως επίσης και το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και καλωσορίζουμε και την διαφάνεια με την οποία προχωράει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπλέον, συμφωνούμε με την δήλωση του Μισελ Μπαρνιέ στην ομιλία του στην Φλωρεντία ότι τα 4-5 εκατομμύρια πολίτες που επηρεάζονται θα πρέπει να συνεχίσουν να ζουν τις ζωές τους σαν να μην είχε συμβεί το Brexit. Γι' αυτό ζητάμε και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο να τηρήσει τις βασικές μας αρχές στις διαπραγματεύσεις και στις επαφές τους ε, με τις δύο κατηγορίες πολιτών. Θεωρούμε ότι η θέση του Ηνωμένου Βασιλείου είναι πάρα πολύ κοντά στις ε, αρχές μας ε, υπό την αίρεση κάποιων διατάξεων για το πεδίο εφαρμογής. Αυτά θα τα εκθέσουμε σε ένα έγγραφο που θα αποστείλουμε προσεχώς στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Ζητάμε λοιπόν ε, η εγγύηση να είναι προτεραιότητα στις διαπραγματεύσεις του άρθρου 50 και να επιβεβαιωθεί αμέσως μετά. Έτσι ώστε οι πολίτες αυτοί να έχουν ε, την βεβαιότητα ότι θα μπορούν να συνεχίσουν τις ζωές τους. Καλώς ορίζουμε λοιπόν την θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συμφωνούμε πως θα πρέπει η εγγύηση αυτή να επιβεβαιωθεί και στην ε, συμφωνία απόσυρσης του Ηνωμένου Βασιλείου για να έχει το καθεστώς ε, διεθνούς δικαίου. Δυστυχώς όμως ε, βλέπουμε μια σοβαρή παράληψη. Φοβόμαστε το τι θα συμβεί στην περίπτωση που δεν επιτευχθεί κάποια συμφωνία. Για τον λόγο αυτό μαζί με τα 3 εκατομμύρια θεωρούμε ότι πρέπει να περιφρουρηθούν τα δικαιώματά μας έτσι ώστε η τελική συμφωνία να μην εξαρτάται από την γενική συμφωνία και να υπάρξει και στην περίπτωση που δεν υπάρξει κάποια συμφωνία. Αλλιώς δεν θα μπορούμε να κοιμηθούμε ησυχοί και κατά την άποψή μας θα συνεχίσουμε να είμαστε διαπραγματευτικά χαρτιά. Με αυτά ως δεδομένο αναμένουμε τώρα την απάντηση του Ηνωμένου Βασιλείου για το εάν η πρόταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα επιβεβαιωθεί βεβαίως στην τελική συμφωνία και αυτό θα εξαρτηθεί από το πώς θα αντιδράσει η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου. Και ζητάμε από την Επιτροπή Αναφορών να μας στηρίξει στην επίτευξη των στόχων που έχουμε τονίσει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you for your... Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέμβασή σας είναι σίγουρα μεγάλη προτεραιότητα για αυτήν την Επιτροπή. Όλη αυτή η εκδήλωση σήμερα είναι αφιερωμένη ε, σε αυτό, έτσι ώστε να συλλέξουμε στοιχεία, μαρτυρίες όπως η δική σας. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ. Ε, δυστυχώς τελειώνει ο χρόνος. Θα δώσω το λόγο για σύντομες παρεμβάσεις ε, πρώτα στην κυρία Ward. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε όλοι οι αναφέροντες. Ευχαριστώ πολύ για αυτά που κάνετε. Ε, χρειάστηκε να παρατήσετε ό,τι κάνατε τον τελευταίο χρόνο έτσι ώστε να πολεμήσετε για τα δικαιώματά σας και θαυμάζω αυτό που κάνετε. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε αυτή τη σχέση μαζί σας. Ε, να σας πω ότι συνεργάζομαι με τους New Europeans για ένα ερωτηματολόγιο και προσπαθούμε να, διασφαλίσουμε τα, να διασφαλίσουμε τα δικαιώματα των πολιτών ανεξάρτητα από τις αποφάσεις της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου. Προσπαθούμε να σταματήσουμε τη μεταχείριση των ανθρώπων ως χαρτί σε μια διαπραγμάτευση και καλούμε την Ευρώπη των 27 να κάνει το σωστό ε, ακόμα και αν η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου κάνει το αντίθετο. Να ξέρετε ότι συνεργάζομαι με τον Ρότζερ Κασάλλας και με τους New Europeans γι' αυτό ε, και αυτό το έγγραφο προτεραιότητας υπεγράφει από 26 ευρωβουλευτές ε, που ανήκουν σε διαφορετικές πολιτικές ομάδες, σε διαφορετικά κράτη-μέλη. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ε, που θα κληθεί να απαντήσει και να δημοσιευτούν τα στοιχεία. Αν θέλετε λοιπόν να μάθετε περισσότερα για την πρωτοβουλία, και να πω εδώ ότι πρέπει ο καθένας μας να κάνει ό,τι μπορεί, όπου μπορεί. Η Επιτροπή Αναφορών είναι πολύ σημαντικό κομμάτι της δουλειάς μας, αλλά πρέπει να την ε, ξεπεράσουμε, να κάνουμε κι άλλα. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Χάνιμπολ έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ όλες τις ε, ομάδες πολιτών που ήρθαν όλες τις πολιτικέ ομάδε Βλέπετε υπάρχουν κάποιοι ευρωβουλευτέ από το Ηνωμένο Βασίλειο. Ε, παίρνουμε την ε, υπόθεση αυτή στα σοβαρά. Κανείς από εμά δεν ήθελε να δει αυτές τις εξελίξεις, αλλά τώρα που έγιναν είναι πολύ σημαντικό εμείς να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Έτσι ώστε οι Ευρωπαίοι πολίτε που ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο και οι Βρετανοί πολίτε που ζουν στην Ένωση να μην δουν αλλάζει καθόλου η ζωή τους, να μην αλλάξουν τα δικαιώματά τους. Εγώ ε, δρεύω στο Λονδίνο και πώς γνωρίζετε η πλειοψηφία των πολιτών της Ένωσης που ζει στο Ηνωμένο Βασίλειο ζει στο Λονδίνο και ως Ευρωβουλευτής του Λονδίνου έχω τεράστια ευθύνη, νιώθω. Ε, πραγματικά, είστε άνθρωποι και όχι πιόνια. Δεν πρέπει να ε, έχετε τέτοια μεταχείριση. Αλλά μην ξεχνάτε ότι το Λονδίνο και η οικονομία και στη χώρα και στην πόλη στηρίζεται σε εσά. Και να είστε σίγουροι πως ε, πολλοί ε, επιφανείς πολιτικοί, ο Δήμαρχος του Λονδίνου για παράδειγμα, το γνωρίζουν αυτό. Εμείς λοιπόν θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Ευχαριστώ πολύ. Να σας ενημερώσω ότι βρίσκεται εδώ στην αίθουσα και εκπρόσωπος της μόνιμης αντιπροσωπείας του Ηνωμένου Βασιλείου και να γνωρίζετε ότι σημειώνουν όλα όσα λέτε, σημειώνουν και ε, τη, τα αποτελέσματα της μελέτης που παρουσιάσαμε και θα την μεταβιβάσουν και στους άλλους συναδέλφους. Νομίζω πως εδώ ήρθε η ώρα να ολοκληρωθεί η πρωινή συνεδρίαση ή όχι. Όχι, πρέπει να συνεχίσουμε. Ωραία, θα ήθελα λοιπόν να συνεχίσω με την αναφορά 847 του Άλαν Μπρέκμαν, ο οποίος όμως δεν είναι παρόν. Βέβαια, εμείς ε, λαμβάνουμε υπόψη όλες τις αναφορές. Έχουμε την ε, αναφορά 955 της κ. Λανχάους ε, από, την, από μια ένωση στη Γαλλία που υπερασπίζεται τα δικαιώματα των Ευρωπαίων Βρετανών πολιτών που ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας δίνω αμέσως το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μας δίνετε τη δυνατότητα να παρουσιάσουμε την αναφορά μας έχει κυλήσει πολύ νερό στα βλάκια από τότε που υποβάλαμε την αναφορά μας και πόσο μάλλον τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Ωστόσο η θέση μας παραμένει η ίδια. Θέλουμε να υπερασπιστούμε τους ε, Βρετανούς πολίτες που διαμένουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους ε, πολίτες ένας που διαμένουν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η συντηρητική κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου έχει καταστήσει επανειλημμένα σαφέ ότι δεν θα δώσει καμία εγγύηση στους Ευρωπαίους πολίτες που ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι να δοθούν αντίστοιχε εγγύησει από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τους Βρετανούς πολίτες που ζουν στην Ένωση. Και ε, αμέσως μετά το Βρετανικό δημοψήφισμα του Ιουνίου του 2016 ε, λένε πως ε, το ενδιαφέρον ε, και κύριο μέλημά τους είναι να προστατεύσουν εμπιστευτεί δηλαδή, τους πολίτες που ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό πρέπει να κάνουν και οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι μας. Η... Το έγγραφο θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφέρει τις κύριες αρχές ε, για την έναρξη διαπραγμάτευση και το έγγραφο της 20ης Ιουνίου 2017 αναφέρει την πορεία των διαπραγματεύσεων που θα οδηγήσουν στη Γενική Συμφωνία. Ωστόσο, το κύριο μέλημά μας ε, είναι να δούμε την κατάσταση όσων Βρετανών ζουν στην ε, Βόρεια Γαλλία. Η κατάσταση διαφέρει σε άλλε χώρε, σε άλλα κρατημέλη. Στη Νότια Ισπανία, για παράδειγμα, δεν είναι διαφορετικά τα πράγματα. Οι Βρετανοί πολίτε είναι κυρίω συνταξιούχοι. Στην Βρετανία, οι Ευρωπαίοι πολίτε είναι ε, νέοι επαγγελματίε. Ενώ στην Γαλλία υπάρχει μία μίξη συνταξιούχων, εργαζόμενων και ανθρώπων οι οποίοι απλά επέλεξαν τη Γαλλία για το ε, του. τους το Βρετανικό Κοινοβούλιο έχει δείξει πλήρη άγνοια για τις ε, ανάγκες ε, των ε, Βρετανών πολιτών στο εξωτερικό. Κανείς δεν έχει σκεφτεί αυτούς τους πολίτες. Για παράδειγμα, ε, ασφάλεια, ιατροφωνικευτική περίθαλψη. Θα παρουσιαστεί ένα νέο πρόβλημα για τους Βρετανούς πολίτες που ταξιδεύουν στην Ευρώπη. Θα είναι πολύ πιο, πολύ πιο δαπανηρό, θα είναι πολύ πιο ακριβό να έχουν ε, φτική περίθαλψη πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ασφαλιστικό σύστημα στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι υποπίεση. Το κόστος των ε, Βρετανών που ζουν στην Ευρώπη ανάρχεται στα 500 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο και υπάρχουν πολλά άλλα τα θέματα. Υπάρχουν θέματα ιδιοκτησίας, ε, εκπαίδευσης, ε, υπηκότητας, υπάρχουν θέματα συντάξεων, μισθών, ε, τραπεζικά ζητήματα, φορολογικά ζητήματα, ασφάλεια ζωής, δικαίωμα στην ελλείψη επιδόματος, ασφαλιστική κάλυψη, κάρτα παραμονής διπλώματα οδήγηση, πάρα, πολλά, ε, πάρα πολλές ε, τι θα γίνει με τι χρεώσει περιαγωγή όταν ε, το Ηνωμένο Βασιλείο αποχωρήσει, με δασμούς τελωνιακού, φορολογία. Καταλαβαίνουμε ότι αυτά είναι αρμοδιότητα της βρετανική κυβέρνησης και όχι της Ευρωπαϊκής Ένωση, όμως για μας πρέπει να αντιμετωπιστούν ως δέσμοι μέτρων, διότι το θέμα αυτό μας καίει. Σας ευχαριστώ πολύ. Επόμενη αναφορά, 808, θα εξεταστεί το απόγευμα. Και η αναφορά 1330 από τον Jeffrey Owen Steele Morgan, ε, ο οποίος λείπει, θα ε, σημειωθεί πως ε, αναφέρεται στην μεστία διάταξη. Νομίζω πως εδώ έχουμε φτάσει στο τέλος της πρωινής συνεδρίασης. Ελπίζω να φάτε καλά γιατί δουλέψατε σκληρά. Και σας ευχαριστώ που ήρθατε εδώ, μας ε, διαφωτίσατε και μας ε, κάνατε νομίζω πιο αποφασισμένους να σταθούμε πλάι σας ε, στο μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ ιδιαίτερα την κυρία Σπαβέντα η οποία μας έδωσε πολύτιμες πληροφορίες.